Dear colleagues, it is uh, time to start also because we here... Είναι καιρός να ξεκινήσουμε αγαπητοί συνάδελφοι και γιατί είναι εδώ ο κύριος ε, Σεύκοβιτς, αντιπρόεδρος ε, που θέλει να μιλήσει και γνωρίζω ότι τα μέλη της Επιτροπής μας θέλουν να τον ακούσουν και να του υποβάλουν ερωτήσεις. Ας μην καθυστερούμε λοιπόν άλλο. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι καταρχάς από του σημείου 1 έγκριση της μεσής διάταξης αν δεν υπάρχουν διαφωνίες μπορούμε να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη έχει. Σημείο 2 να σας πω ότι έχουμε σε 20 γλώσσες σήμερα διερμηνία και όσοι ήθιστε ο φάκελος με τα θέματα της σημερινής συνεδρίασης διατίθεται ηλεκτρονικά. Η συνεδρίασή μας μεταδίδεται στο διαδίκτυο. Τρίτο σημείο ανακοινώσεις του Πρόεδρου σχετικά με τις συστάσεις των συντονιστών. Σας τις διαβιβάσαμε ηλεκτρονικά και αν δεν έχετε αντίρρηση θεωρούμε ότι εγκρίνονται. Τέταρτο σημείο. Και φτάνουμε στο δικό σας ε, σημείο. Θα πρέπει να σας ενημερώσω για τις τρέχουσες διοργανικές διαπραγματεύσει. Έγινε ο τέταρτος τριμερής διάλογο για τα νέα τρόφιμα Και έχουμε διαφωνίε με την Κομισιόν και το Συμβούλιο για δύο σημεία κυρίω. Δηλαδή, πρώτον, κατ' εξουσιοδότηση πράξη, γιατί εμεί εμένουμε στην άποψή μα. Και το δεύτερο θέμα είναι η κλωνοποίηση. Δεν έχουμε την ίδια θέση με το Συμβούλιο Εμείς τελείσαμε άρθρο, το Συμβούλιο δέχεται να μας παραχωρήσει αιτιολογική σκέψη. Πάντως έχουμε υποβάλει την τελική μας πρόταση στο Συμβούλιο για το ενδεχόμενο μιας συμφωνίας και περιμένουμε την απάντησή του, την οποία και αναμένουμε στα τέλη αυτής της εβδομάδας για το όλο πακέτο. Και έπειτα Φτάνουμε στο σημείο 5 της Μεσής Διάταξης, ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τον Αντιπρόεδρο Σεύκοβιτς. Στα πλαίσια του δεδομένου διαλόγου που έχουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως συνηθίζω θα δώσω αμέσως το λόγο στον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που είναι αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση για να μας κάνει την παρουσίασή του και θα ακολουθήσει πάλι ως ήθιστε ανταλλαγή απόψε και ερωταπαντήσεις. Μας ενδιαφέρουν ορισμένα συγκεκριμένα σημεία της θεματολογίου σας. Παρακολουθούμε τις διαπραγματεύσεις εν ώψη της διάσκεψης COP21 στο Παρίσι το Δεκέμβρη και μας ενδιαφέρει πραγματικά να ακούσουμε τις προτεραιότητές σας αλλά και τις εξελίξεις, πώς προχωρούν διαπραγματεύσεις και τι άλλο έχετε να μας πείτε για τα θέματα που άπτωτε του χαρτοφυλακίου σας, ενεργειακή ένωση, απαλλαγή από τον άνθρακα κτλ. Τα μέλη της Επιτροπής μας και όλοι οι υπόλοιποι θέλουν να ακούσουν τις τελευταίες ειδήσει και σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα εργασίας του 2015 και το πρόγραμμα εργασίας 2016 που θα το συζητήσουμε προσεχώς με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έχετε το λόγο και 15 λεπτά στη διάθεσή σας για να μας παρουσιάσετε τις δικές σας προτεραιότητες σε σχέση με τα θέματα αυτά και για το βασικό ζήτημα που μας απασχολεί σήμερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε Λαβία, αξιότιμα μέλη της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι. Ε, ήταν στο ημερολόγιο μου ότι πότε συναντηθήκαμε την περασμένη φορά, την τελευταία φορά. Δεν ήταν και πριν από πολύ καιρό, ήταν περίπου πριν από τέσσερις μήνες. Τότε σας είχα παρουσιάσει ένα όραμα για μια φιλόδοξη ενεργειακή ένωση και συζητήσαμε και είπαμε γιατί ήταν σημαντικό οι Ευρωπαίοι να έχουν προσιτή, ασφαλή, ανταγωνιστική και βιώσιμη ενέργεια και τότε είχα και την ευκαιρία να ακούσω εσάς τις ιδέες σας και είδατε ότι πολλές από τις ιδέες σας συμπεριλήφθησαν στο τελικό σχέδιο της δημοσίευσης για την Ενεργειακή Ένωση που ε, παρουσιάστηκε τέλος Φεβρουαρίου. Πρόκειται για μια ανακοίνωση που μετέφραζε το όραμα που συζητήσαμε την περασμένη φορά σε συγκεκριμένη στρατηγική. Λίγο μετά την παρουσίασή της, η Στρατηγική για την Ενεργειακή Ένωση υιοθετήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, καλωσορίστηκε θερμά από πολλές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και νομίζω ότι έγινε πολύ καλά ε, αποδεκτή από τους πολίτες και μεγάλους εμπλεκομένους. Όμως η στρατηγική αυτή είναι μόνο η αρχή μιας πολύ αποφασιστικής θα έλεγα διαδικασίας. Τώρα ήρθε η ώρα να υλοποιήσουμε τα ωφέλη της Ενεργειακής Ένωσης ήρθε η ώρα να περάσουμε από τα λόγια στα έργα. Σήμερα το πρωί ανακοίνωσα μια νέα και κρίσιμη φάση, δηλαδή τη, τη φάση της εφαρμογής μέσα από σειρά συγκεκριμένων δράσεων σε πολιτικό, διπλωματικό και νομοθετικό επίπεδο. Όπως και στην προηγούμενη φάση θα φροντίσω να είναι κοινή προσπάθεια που θα προωθηθεί από όλους τους επιτρόπους που ανήκουν στην οικογένεια της Ενεργειακής Ένωσης και σε στενή συνεργασία βέβαια και με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Χρειαζόμαστε ε, μια συλλογική προσέγγιση γιατί απεδείχθη αυτή πολύ επιτυχής. Πολύ γρήγορα να καλύψω τα τρία αυτά σκέλη. Πρώτα το πολιτικό. Νομίζω ότι είναι σαφές ότι τώρα θα πρέπει η Ενεργειακή Ένωση να πάει στα κράτη-μέλη, δηλαδή στα εθνικά κοινοβούλια, στους δημάρχους, στους κοινωνικούς εταίρους, στους εκπροσώπους των επιχειρήσεων, τους φοιτητές, στα think tanks, σε ομάδες προβληματισμού. Αυτή, αυτός είναι ο στόχος της περιοδίας Ενεργειακής Ένωσης που ανέφερα όταν την ανακοίνωσα νωρίτερα σήμερα. Να εξηγήσουμε επιτόπου δηλαδή ότι η Ενεργειακή Ένωση συνεπάγεται τριπλό κέρδο επειδή ωφελεί καταναλωτέ, την οικονομία και το περιβάλλον. Επίσης θα πρέπει να μας δώσει μια ευκαιρία να συζητήσουμε με τους πολίτες και τους πολιτικούς παράγοντες τι σημαίνει η Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Ένωση για την κάθε χώρα χωριστά. Ε, επίσης, κατά τις επισκέψεις στις χώρες θα εντοπίσω τις βέλτιστες πρακτικές, τα χαρακτηριστικά παραδείγματα σε όλη την Ευρώπη για το πώς θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε αυτή τη βαθιά ε, ενεργειακή μετάβαση που χρειάζεται η Ευρώπη. Ε, είναι πολύ σημαντικό να αξιοποιήσουμε τη γνώση, την πρακτική εμπειρία των τοπικών παραγόντων, δημάρχων, ΜΜΕ, επενδυτών. Θα πρέπει όλα αυτά να τα κάνουμε πιο γνωστά, να τα αναδείξουμε αλλά και να τα προωθήσουμε. Ε, χρειάζονται όλοι αυτοί ε, όθηση από εμά που λαμβάνουμε τις αποφάσεις. Η περιοδία της Ενεργειακής Ένωσης θα επιτρέψει στις εθνικές κυβερνήσεις να αξιολογήσουν από την πλευρά τους τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις στην ενέργεια και το κλίμα και να συμπληρώσουν την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να δώσουν και πληροφορίες πρόσθετες. Ο Εθνικός Διάλογος θα καταλήξει σε φακέλους ειδικού για κάθε χώρα. Και όταν πάρουν την τελική τους μορφή αυτοί οι φάκελοι και οι συστάσεις θα κοινοποιηθούν και θα αποτελέσουν μέρος της πρώτης κατάστασης της Ενεργειακής Ένωσης που θα εγκρίνουμε το φθινόπωρο. Χρειαζόμαστε ένα ισχυρό, δυναμικό, ολοκληρωμένο, χωρίς αποκλεισμούς, εξυμφρονισμένο σύστημα διακυβέρνηση για την Ενεργειακή Ένωση. Φιλοδοξώ να κάνω την κατάσταση για την Ενεργειακή Ένωση ένα μέσο ισχυρό που θα παρακολουθεί την πρόοδο και θα εντοπίζει ένα απομείναντα εμπόδιο, όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο όπως εξήγησα, αλλά και σε περιφερειακό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αυτό το μέσο δεν θα ετοιμαστεί απομονωμένο στις Βρυξέλλες, μακριά από τις πραγματικές προκλήσεις υλοποίησης για να είναι αποτελεσματικό θα χρειαστεί τα κράτη-μέλη να το θεωρήσουν δικό τους σε πολιτικό επίπεδο. Το ίδιο και οι παράγοντες επιτόπου, οι ε, ρυθμιστικές αρχές, οι κοινωνικοί εταίροι, οι δήμαρχοι, οι επιχειρήσεις κλπ. Στόχος μου λοιπόν είναι ήδη από τώρα να εγκαθιδρύσω τακτικό διάλογο μαζί τους. Θα χρειαστεί είμαι σίγουρο στα επόμενα χρόνια. Αυτό το ισχυρό σύστημα διακυβέρνηση θα ενισχύσει την συνοχή των δράσεων της Ενεργειακής Ένωσης και το συντονισμό, την παρακολούθηση, εποπτεία και πίεση από τους ομολόγους από την πλευρά των κρατών μελών. Για να διευκολύνουμε το έργο αυτό θα εξυγχρονίσουμε και τις πολλές υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων. Όταν άρχισα να καταγράφω πόσες υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων ε, υπάρχουν σε επίπεδο κρατών μελών, έφτασα στον αριθμό των 200. 200 διαφορετικές εκθέσεις που πρέπει να αποστέλλονται από τα κράτη-μέλη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, θέλουμε να αλλάξουμε το σύστημα και με αυτό κατά νου θα προτείνουμε κάθε κράτος μέλος να έχει ένα ενιαίο πρόγραμμα ενέργειας και κλίματος, εθνικό πρόγραμμα το οποίο θα καλύπτει τα βασικά στοιχεία της Ενεργειακής Ένωσης. Βεβαίως η δημοκρατική διάσταση είναι εδώ το κλειδί. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσει να εμπλέκεται σε όλο αυτό το ταξίδι. Ξαναγυρίζω στην ε, περιοδία της Ενεργειακής Ένωσης ε, για λίγο. Ελπίζω ότι εσείς, τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, θα με βοηθήσετε να φέρω την Ενεργειακή Ένωση στους πολίτες, σε κάθε εκλογική σας περιφέρεια. Κάποιοι από εσάς ήδη εκφράσατε ενδιαφέρον να έρθετε μαζί μου και να συμμετέχετε σε αυτή τη δημόσια συζήτηση. Αυτό το χαιρετίζω και καλωσορίζω την ευκαιρία ε, για να απευθύνω πρόσκληση σε όσους από σας ενδιαφέρονται για να συμμετέχουν. Ε, στο τέλος αυτής της περιοδίας θα υποβάλω την πρώτη κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα συζητήσουμε μαζί. Ε, επειδή αυτή, αυτό το στρατηγικό έγγραφο θα είναι η αρχή μιας δυναμικής διαδικασίας όπου τα κράτη-μέλη θα υποβάλουν ε, τακτικά αναφορές για την πρόοδο προς την Ενεργειακή Ένωση, είναι σημαντικό να έχουμε συνεκτική πολιτική συζήτηση. Ε, θα συνεργαστούμε ούτως ώστε να βελτιώσουμε την πολιτική δέσμευση των κρατών μελών υπέρ της Ενεργειακής Ένωσης. Επίσης, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο γενικά και η Επιτροπή σας ιδιαίτερα θα είναι στρατηγικός εταίρος σε όλες τις δέσμες του νομοθετικού πολιτικών μέτρων που προετοιμάζονται. Εκτός από το πολιτικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή to touch upon. And here we clearly have a double... ε, όχι. Ε, εκτός από το πολιτικό σκέλος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα... COP21 in Paris. And secondly... Υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα και εμπλοκή καναλιών. Χρειάζεται και ενεργειακή διπλωματία. Θα συμφωνήσετε ότι σε λίγους μήνες θα έχουμε ιστορική ευκαιρία να αντιμετωπίσουμε την κλιματική αλλαγή σε διεθνές επίπεδο. Οι δράσεις μας στην Ευρώπη είναι αποτελεσματικές μόνο αν αποτελέσουν μέρος μιας γνήσιας παγκόσμιας προσπάθειας. Πολλά μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τώρα ε, δίνουν μάχη υπέρ αυτής της υπόθεσης όταν συναντούνται με εθνικούς ε, ηγέτες. Η Αντιπρόεδρος Μογκερίνη, ο Επίτροπος Άριας Κανέτε, ε, ο βασικός διαπραγματευτής, ο Επίτροπος Μιμίκα και άλλοι επίτροποι συμμετέχουν σε αυτή την κοινή προσπάθεια στα πλαίσια της COP21. Και ξέρω ότι το, η αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου επίσης μας βοηθεί να μιλούμε με μία φωνή ε, ως Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτό το σημαντικό θέμα. Εγώ θα αρχίσω έναν διάλογο, θα συμμετάσχω σε διάλογο με κάποιους Αφρικανούς εταίρους. Αρχίσαμε συζήτηση με τον εκπρόσωπο της Επιτροπής της Αφρικανικής Ένωσης ε, όταν ήρθαν στις Βρυξέλλες την περασμένη φορά και επίσης έχουμε και κάποιες δραστηριότητες εξάπλωσης των προγραμμάτων μας στην Αφρική σε στενή συνεργασία και συντονισμό με το Γαλλική Προεδρία COP21. Ε, ένα άλλο θέμα αφορά τις ανάγκες της ε, ε, Ευρώπης και τη βούλησή της να διαφοροποιήσει τις ε, πηγές ενέργειας, τους προμηθευτές, τις ε, περιοδίες, ε, τις διαδρομές που ακολουθεί η ενέργεια. Ο Επίτροπος Αρίας επίσης πήγε σε χώρες της Βορείας Αφρικής. Επίσης συζητούμε με τη Ρωσία για την εφαρμογή του χειμερινού πακέτου και συνεργάστηκα με εταίρους για να προχωρήσει ο νότιος διάδρομος που θα φέρει φυσικό αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη. Και βεβαίως αυτό το έργο θα συνεχιστεί διότι είναι τεράστιο έργο και πρέπει να ολοκληρωθεί. Επίσης ε, συνεργαζόμεθα με τον Επίτροπο Αρία Κανέτε για να βεβαιωθούμε ότι η Νοτιοανατολική Ευρώπη επιτέλους θα ενταχθεί στα ενεργειακά συστήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και κάθε χώρα από αυτή την περιοχή θα μπορεί να προμηθεύεται αέριο από ε, τουλάχιστον τρεις διαφορετικές πηγές για να ε, ξεπεράσουμε την ενεργειακή απομόνωση των χωρών για τόσα χρόνια. Τέλος κύριε Πρόεδρε το τρίτο επίπεδο εκτός και παράλληλα με το πολιτικό και το διπλωματικό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εργάζεται σκληρά για να παρουσιάσει σειρά νομοθετικών και άλλων πρωτοβουλειών που καλύπτουν και τις πέντε διαστάσεις της Ενεργειακής Ένωσης. Εγκρίνοντα όλε τι πρωτοβουλίε, ο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ω συνομοθέτη θα είναι θεμελιώδη. Πολύ σύντομα να παρουσιάσω τι βασικέ προτάσει που θα υποβάλει η Επιτροπή φέτος πολύ γρήγορα να αναφερθώ στις πέντε διαφορετικές διαστάσεις. Τομέα ασφάλεια εφοδιασμού. Μέχρι το τέλος του έτους θα παρουσιάσουμε μια πρόταση για την αναθεώρηση της ασφάλειας του αερίου, του ε, κανονισμού για τον εφοδιασμό, να διασφαλίσουμε τους ε, εφοδιασμούς σε περίπτωση ε, διαταραχής, να ενισχύσουμε την συνεργασία σε περιφερειακό επίπεδο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να βελτιώσουμε την αντιμετώπιση της κρίσης. Θα χρειαστεί μεγαλύτερη διαφάνεια στη συμβάση για το αέριο με, με τρίτα μέρη, όπως προβλέπει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Μαρτίου. Ε, επίσης στρατηγική για το υγρό υγραέριο και την αποθήκευση. Η αναθεώρηση της απόφασης για τις διακυβερνητικές συμφωνίες προβλέπεται για του χρόνου. Ε, για την εσωτερική αγορά το Φεβρουάριο ο Επίτροπος Αρίας Κανιέτε παρουσίασε ανακοίνωση για το πώς θα φτάσουμε στο στόχο διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας 10%. Ε, εκτός από ε, ε, την διασυνδεδεμένη υποδομή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα γίνει πραγματικότητα εκτός και αν έχουμε μια πραγματική εσωτερική αγορά όπου θα εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να φροντίζει ότι το ενωσιακό δίκαιο θα εφαρμόζεται σωστά και θα επιβάλλεται και θα χρησιμοποιήσει τις διαδικασίες επί παραβάση αν χρειαστεί. Επίσης θα κάνουμε ε, μία ε, ανακοίνωση σχετικά ε, με τη, το, το, την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το σχεδιασμό της, καλύτερη ολοκλήρωση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενίσχυση του ΑΣΕΡ, ενέργεια που παράγεται από τους καταναλωτές και τις λιανικές αγορές, νέα συμφωνία για τους καταναλωτές. Αυτό θα το ακολουθήσει τον επόμενο χρόνο ε, μια σειρά από φιλόδοξες νομοθετικές προτάσεις. Ε, ενεργειακή ε, απόδοση θα παρουσιάσω με την αναθεώρηση της σχετικής οδηγίας σήμανσης της ενέργειας. Επίσης, μια στρατηγική για την θέρμανση και ψήξη ε, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό γιατί στην κατανάλωση ενέργειας. Μέχρι το τέλος του έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει και ένα κυκλικό πακέτο οικονομικό το οποίο ετοιμάζεται τώρα ε, και συντονίζεται από τον Αντιπρόεδρο Κατάινεν. Θέλουμε να ε, μην λάβουμε μόνο υπόψη μας την, την, τη σπατάλη ενέργειας αλλά να κλείσουμε και το βρόχο ε, συμπεριλαμβάνοντας ε, για παράδειγμα και το σχεδιασμό προϊόντος. Για την απαλλαγή από ανθρακούχες ε, εκπομπές θέλω να σας ευχαριστήσω για την συμφωνία επί του αποθέματος σταθερότητας στην αγορά και τώρα, γιατί έτσι μπορούμε τώρα, να υποβάλλουμε πρόταση για την αναθεώρηση του συστήματος ETS, δηλαδή το σύστημα εμπορίας εκπομπών, ως τμήμα του, του, της νομοθετικής δέσμης του καλοκαιριού. Αυτό είναι σημαντικό για να ε, ρυθμίσουμε την αγορά άνθρακα. Επίσης θέλουμε να γίνουμε υπαριθμόν ένα στις, ανα, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ε, το προπαρασκευαστικό έργο τώρα θα οδηγήσει το 2016-2017 σε φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Το νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να δώσει ασφάλεια και βεβαιότητα στους επενδυτές σχετικά με την χρήση των ανανεώσιμων σε όλα τα επίπεδα. Ε, έρευνα καινοτομία. Για να παραμείνουμε ηγέτες στον τομέα αυτό πρέπει να, έχουμε να διατηρήσουμε ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Το ανανεωμένο πρόγραμμα δράσης για τη στρατηγική ενεργειακή τεχνολογία που θα δημοσιευθεί το Σεπτέμβριο θα κάνει μια ανάλυση του τεχνολογικού τοπίου και τις δράσεις που πρέπει να ληφθούν. Λίγο μετά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα προτείνει την ε, παγκόσμια τεχνολογική ε, πρωτοβουλία ηγετικής θέσης που θα εστιάζεται σε νέες τεχνολογίες στην ενέργεια και το κλίμα. Ε, οπωσδήποτε θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει ομαδικό πνεύμα και συλλογική προσπάθεια ούτω ώστε η στρατηγική της Ενεργειακής ε, Ένωσης να ολοκληρωθεί γρήγορα. Έχω οργανώσει στοχευμένες συναντήσεις ε, της Ομάδας Ενεργειακής Ένωσης ούτως ώστε η εργασία να μπει στη σωστή τροχιά. Ε, έχουμε την, ε, το σχεδιασμό της αγοράς, ε, τις λιανικές αγορές, διάφορα άλλα θέματα όπως αέριο, έρευνα και καινοτομία και στα πλαίσια αυτής της συλλογικής προσπάθειας του χρόνου θα μιλήσουμε για ενεργειακή απόδοση, ανανεώσιμα, θέματα που δεν αφορούν την εμπορία εκπομπών και την απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές. Ε, ζητώ συγγνώμη αν μακρηγόρησα, αλλά όπως βλέπετε ε, πολλή δουλειά μας περιμένει ακόμα, αλλά άρχισε ε, πλέον 100% η διαδικασία για την Ενεργειακή Ένωση. Ε, το, η συνάντηση αυτή αποτελεί μέρος του διαρθρωμένου διαλόγου. Να συνοψίσω λοιπόν τα πιο σημαντικά. Ε, για φέτος μόνο ε, επαναλαμβάνω ότι θα υποβάλλουμε ένα πρώτο πακέτο νομοθετικό μέχρι το καλοκαίρι ε, για το νέο σχεδιασμό της αγοράς, τις ελληνικές αγορές, την εμπορία εκπομπών, την σήμανση ενέργειας και τις ανανεώσιμες. Ε, το, θερινό, το χειμερινό πακέτο με συγχωρείτε, θα έχει αναθεωρημένο κανονισμό για την ασφάλεια του εφοδιασμού σε αέριο ε, για το υγραέριο και το δεύτερο κατάλογο PCI. Ε, εν τω μεταξύ θα, έχουμε την, θα, εγκριθεί η κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και όπως είπαμε θέρμανση και ψήξη ως στρατηγική. Ε, πιστεύω ότι και όλοι οι Επίτροποι και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα εργαστούν για να ολοκληρωθούν επιτυχώς οι διαπραγματεύσεις για το κλίμα επίσης. Για το 2016 πρέπει να αναφέρω νομοθετικές προτάσεις για το σχεδιασμό της αγοράς, την ασφάλεια του εφοδιασμού σε ηλεκτρική ενέργεια, το πακέτο για την ενεργειακή, ενεργειακή απόδοση και ενδεχομένως και το, την νομοθετική δέσμη για την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε για το ενδιαφέρον σας, για την υποστήριξή σας. Προσβλέπω στη συνέχιση της συνεργασίας μας επί αυτών των πολιτικών, νομοθετικών και διπλωματικών μετόπων και επειδή σας ανέφερα ενδελεχώς ε, τα τρία διαφορετικά σκέλη ε, δράσης μας, περιμένω τις, ε, τα σχόλιά σας επί όλων αυτών. Εγώ σας ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος. Τώρα θα ξεκινήσουμε δίνοντας το λόγο πρώτα στους συντονιστές μας. Να μην ε, λησμονείτε ότι δεν πρέπει να ξεπερνάει ο καθένας σας τα δύο λεπτά. Ο Πίτερ Λίζερ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Νομίζω ότι ήταν πολύ ενθαρρυντικά αυτά που μας είπατε για την Ενεργειακή Ένωση. Θέλω να υπογραμμίσω ιδιαίτερα ότι και εσείς θα αναδείξατε ιδιαίτερα το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Για πρώτη φορά το άκουσα σήμερα τόσο καθαρά να λέγεται ότι σε αυτούς τους τομείς όπου μέχρι τώρα υπήρχαν αποφάσεις και συναπόφαση ε, θα έχουμε και νέα πρόταση για οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είναι πολύ ωραίο και το θέμα της ε, διακυβέρνησης ε, όπου έπαιζε, έπαιζε λιγότερο ρόλο, μικρότερο ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το θέμα λύθηκε και είναι καλό. Θα ήθελα να επιβεβαιώσετε παρακαλώ ότι θα υπάρξει και νέα πρόταση οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση ε, μέχρι το 2020. Θα ήθελα να μου το πείτε αυτό. Επίσης, σε αυτά τα πλαίσια υπάρχει μια αναντιστοιχία στο κείμενο για την Ενεργειακή Ένωση όπως παρουσιάστηκε. Η ενεργειακή απόδοση εκεί αναφέρεται ε, στο 27% κάποια άλλη στιγμή 30% αλλά ο πρόεδρος Γιούνκερ είχε πει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι το 30% το θέτει ως ελάχιστο στόχο. Γι' αυτό θα πρέπει να μας εξηγήσετε πώς ε, αυτή την υποχρέωση που ανέλαβε ο Ζαν Κλοντ Juncker θα την εφαρμόσει στην πράξη. Τέλος, το Energy Labeling και σχετική οδηγία ε, υπήρχε και στην ημερήσια διάταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τώρα το αναφέρεται για τον Ιούλιο. Το λέτε ότι θα γίνει τον Ιούλιο. Γιατί δεν υπευλήθη σχετική πρόταση ε, τον περασμένο μήνα όπως είχε αρχικά σχεδιαστεί. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον Ματία Σκρότη για τους σοσιαλιστές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Ο πυρήνας της ε, ενεργειακής πολιτικής που μας συνδέει και σε αυτό είναι το θέμα του συστήματος ε, εμπορίας εκπομπών αυτό είναι ένα οικοδόμημα στο οποίο εργαζόμεθα όλοι. Το απόθεμα της αγοράς ενέργειας επίσης ε, κατέληξε σε συμφωνία με το Συμβούλιο. Μπορεί αυτό να επιβεβαιωθεί, αλλά εμείς ε, ε, ασκήσαμε πιέσεις γιατί θέλαμε αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας των εκπομπών πριν από το καλοκαίρι του 2015. Αυτά τα λέγαμε συχνά. Υποθέτω ότι το 2015 λοιπόν θα προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα και είμαι πεπισμένος ότι όλοι οι συμμετέχοντες και όλοι οι πιθανοί επενδυτές ε, παρακολουθούν την Ενεργειακή Ένωση και θέλουν βεβαίως σαφείς προϋποθέσεις πλαίσιο. Περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον όλοι την πρόταση, τι μορφή θα έχει και βέβαια τι θέση θα πάρουν τα διάφορα λόμπι εις ό,τι αφορά την ε, διαρροή άνθρακα για παράδειγμα πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το, πώς συζητήθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα με ενδιαφέρε να ξέρω αυτό δηλαδή θα πρέπει εδώ να ε, έχουμε διατηρήσει, να διατηρήσουμε ανοιχτές τις πύλες ή μήπως το 2008 και το 2009 είμαστε υπερβολικά γενναιόδοροι σχετικά με την αντιμετώπιση του carbon leakage της διαρροής ε, άνθρακα ε, και την ε, κοινή αυτή, το κοινό σύστημα που είχαμε και που οδήγησε σε πάρα πολλές άδειες. Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει να τα βελτιώσουμε κατά την αναθεώρηση για να λειτουργεί το σύστημα και να ε, υπάρχει μια γενικότερη καθοδήγηση. Οι Υπουργοί Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πιστεύω πολύ δημιουργικοί. Ε, νομίζω ότι μπορούν να ε, ρυθμίσουν και πολλά σχετικά θέματα ε, όπως και ε, θέματα φόρου στον τομέα αυτό, ούτως ώστε να προχωρήσει η Ενεργειακή Ένωση. Άλλη ερώτηση, δεύτερη. Ε, με ποια ιδιότητα θα πάμε στο Παρίσι. Υπάρχει ας πούμε το, ένα, ε, ε, μια κοινωτική ενωσιακή ιδιότητα ή τι ρόλο θα παίξουμε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Εμείς θα ετοιμάσουμε έκθεση, όχι μόνο ψήφισμα. Ε, έχουμε δηλαδή ήδη αναθέσει σε συνάδελφο την έκθεση αυτή και μας ενδιαφέρει να ξέρουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα προωθήσει τα θέματα αυτά γιατί στο Παρίσι υπάρχει μεγάλη ευκαιρία. Χρειαζόμαστε μια νομικά δεσμευτική συμφωνία και όχι μόνο γενικόλογες δηλώσεις προθέσεων. Οπότε ε, θέλουμε και σε αυτό κάποια θέματα. Για να μην ε, μακρηγορήσω άλλο, σταματώ εδώ. Ευχαριστώ πολύ από η κυρία Ιβζινεύσκα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ που είσαστε εδώ. Ε, επανειλημμένα έχω παρουσιάσει την αρνητική μου θέση όσον αφορά ε, τις ε, ε, θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά την απαλλαγή από, το, τις εκπομπές άνθρακα. Για μία ακόμα φορά δεν γίνεται λόγος για τα δηληστήρια, τα προϊόντα τους και τα, παρά, τα υποπροϊόντα τους. Ε, ή ε, εάν γίνουν δεκτές όλες οι προτάσεις ε, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τότε θα πρέπει τα δηληστήρια να υπομείνουν ένα πάρα πολύ μεγάλο κόστος ε, ε, και αυτό σημαίνει ότι θα μειωθεί η ανταγωνιστικότητά τους, πράγμα που με τη σειρά του σημαίνει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, θα εξαρτάται όλο και περισσότερο από εξωτερικές πηγές ενέργειας. Όσον αφορά την κλιματική ε, αλλαγή είναι γεγονός ότι και σε αυτό το πλαίσιο ε, χάνει τον ρυθμό της και την ανταγωνιστικότητά της ή ε, την ανταγωνιστικότητά του ο τομέας των δηληστηρίων. Όσον αφορά το αργό πετρέλαιο δεν είναι δυνατόν να λησμονεί κανείς την μεγάλη εξάρτηση των χωρών της Ανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης όσον αφορά την πρώτη ύλη, την εισαγόμενη από τη Ρωσία. 90% ε, των αναγκών της Πολωνίας καλύπτονται με αυτόν τον τρόπο. Επομένως η ασφάλεια του ανεφοδιασμού είναι προβληματική. Ε, ε, χρειαζόμαστε πολύ σαφείς θέσεις και δεσμεύσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Τώρα που δουλεύετε για το τελικό σχήμα της Ενεργειακής Ένωσης θα πρέπει να λάβετε υπόψη φυσικά και την συνέχιση των συμβατικών μορφών ενέργειας όπως είναι το πετρέλαιο ή το φυσικό ε, αέριο. Ε, θα ήθελα να μας πείτε δύο λόγια, τι έχετε προβλέψει για αυτά. Επίσης, ε, όσον αφορά την τελική μορφή της Ενεργειακής Ένωσης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη ε, και τα ζητήματα των κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου. Δεν είναι δυνατόν όλα να, όλες οι μορφές να αντικατασταθούν από πράσινες μορφές ενέργειας. Θα πρέπει βεβαίως βεβαίως να δούμε και άλλους τρόπους διαφοροποίησης ε, του πετρελαίου και του ε, αερίου, αλλά παρόλα αυτά να μην λησμονούμε και αυτές τις μορφές ενέργειας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γερβάν Μπράντι από την, από, από την Ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να γίνει πιο ανταγωνιστική στον κόσμο η δική μας ε, ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι πραγματικά να γίνει μια οικονομία ε, εντελώς απαλλαγμένη ή σχεδόν εντελώς απαλλαγμένη από τις ε, ανθρακούχες εκπομπές. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Επίτροπο ε, για το, τις εισαγωγικέ του παρατηρήσεις και να τον ευχαριστήσω και για την παρουσίαση που μας έκανε όσον αφορά την ενεργειακή του περιοδία ε, σήμερα το πρωί. Ε, εγώ το, βλέπω, το έβλεπα έτσι σαν κάτι πολύ μυστηριώδες αυτή την περιοδία, ίσως και άλλη μεταξύ ημών, αλλά δεν είναι και αστείο τελείω, γιατί νομίζω ότι χρειάζεται μαγεία και μυστήρια κύριο έτσι να κατανοήσουν οι μένες Πολιτείες ε, ότι ε, εμείς δεν εκπροσωπούμε 28 μεμονωμένες ενεργειακές πολιτικές αλλά έχουμε ε, μία ενιαία ενεργειακή ένωση η οποία θα μας δώσει τη δυνατότητα στο μέλλον να έχουμε φτηνή και καθαρή ενέργεια. Έχω κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά αυτήν την περιοδία. Ζητάτε, ρωτάτε τα τα κράτη-μέλη να έχουν ενιαίο κλιματικό ε, πρόγραμμα. Αυτό καταρχήν είναι καλό. Αλλά τους ζητάτε και οδικό χάρτη μέχρι το 2030. Οπότε και θα πρέπει να φτάσουμε σε μια οικονομία με εκπομπές περίπου στο 0% ε, γιατί θα πρέπει ήδη να δουλεύουν πάνω στο θέμα αυτό τα κράτη-μέλη. Και επ' αυτού ε, το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker. Θα συμφωνήσετε μαζί μου ότι ε, κάθε επένδυση που θα συμπεριληφθεί σε αυτό το πρόγραμμα θα πρέπει να βασίζεται ε, σε αυτήν την απαλλαγμένη από άνθρακα οικονομία γιατί διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να προβλέψουμε το τι θα γίνει μετά από 20-30 χρόνια. Τέλος κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ζητήσω από τον Επίτροπο να μου πει το εξής. Ακούω διάφορες φήμες ότι η Κομισιόν ε, έχει αφαιρέσει ε, τις ε, επιδοτήσεις των υδρογονανθράκων και των Um, και των ορυκτών καυσίμων από τον προγραμματισμό. Ε, η Ιταλία ε, ε, πέρσι είχε ζητήσει κάτι αντίστοιχο. Πάντως σύμφωνα με το Διεθνές Ομισματικό Ταμείο εξακολουθούμε να δίνουμε πολλά δις ευρώ όσον αφορά τις επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων. Κάπως θα πρέπει να σταματήσει η πολιτική πολιτική αυτή και να ε, διορθωθούν τα δεινά τα οποία έχει προκαλέσει. Ε, τι γίνεται λοιπόν, συνεχίζεται ε, με τις επιδοτήσεις, τις έχετε σταματήσει, έχει ξεκινήσει το ξεκαθάρισμα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λέει ο Πρόεδρος από την πλευρά της Γουέ κυρία Κονέτσκα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε για τις εισαγωγικέ σας παρατηρήσεις και ευχαριστούμε που μας ε, ε, παρουσιάσατε αυτό το ε, πρόγραμμα. Καλό είναι που έρχεται κάποιος και μας δίνει μια συγκεκριμένη ημερομηνία γιατί πολύ σπάνια ακούμε συγκεκριμένες ημερομηνίες εδώ και επίσης ε, πολύ σπάνια οι ημερομηνίε αυτές ε, έτσι είναι λογικές και εφαρμόσιμες. Θα τις ελέγξουμε και σε τούτη την περίπτωση. Υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα πράγματα σε αυτά που είπατε. Μιλήσατε για την ε, για την διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, αλλά υπάρχει το θέμα της ε, ε, υποδομής. Για να αλλάξουν οι υποδομές θα χρειαστούν πάρα πολλά χρήματα. Πολλές χώρες μπορούν να ανταποκριθούν βεβαίως, αλλά όταν θα έχουμε την υποδομή η οποία θα μπορεί να λειτουργήσει αλλά ε, υπάρχει αυτός ο, ο ενδιάμεσος χρόνος τον οποίο εσείς δεν αναφέρετε στο πρόγραμμά σας. Επομένως θα ήθελα να μου πείτε ε, ποια είναι η άποψή σας όχι μόνο όσον αφορά την διαφοροποίηση ε, και την μείωση των ε, εισαγωγών αλλά τι γίνεται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ας πούμε για την Τσεχική Δημοκρατία η κατάσταση αρχίζει και γίνεται επικίνδυνη. Εάν δεν βελτιώσουμε την υποδομή μας θα έχουμε πρόβλημα. θα εξακολουθεί αν ε, δεν ε, συνεχίσετε να στηρίζετε ε, τις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, τότε κάποια στιγμή οι, υποδομή, οι υποδομές θα έχουν πρόβλημα γιατί δεν θα μπορούν πλέον να αντιμετωπίσουν τη ζήτηση. Δεύτερο, η καταπολέμηση της ενεργειακής φτώχειας. Νομίζω ότι όλο και περισσότεροι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι είτε ήδη βρίσκονται μέσα στην ενεργειακή φτώχεια είτε κινδυνεύουν ε, να βρεθούν ε, στα όρια της, ε, αυτής της ενεργειακής ένδυας. Πολλά πρέπει να γίνουν κατά αυτή την έννοια και θα πρέπει να υπάρξει μια ενιαία λύση. Επομένως, πώς προτίθεστε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα της ενεργειακής ένδυας και έχετε δυνατότητα να εισαγάγετε αυτά τα νέα στοιχεία σε τρεις μήνες. Ευχαριστώ πολύ για τους πράσινους. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Ε, για τις αρκετά λεπτομερείς ε, επεξηγήσεις που μας δώσατε για το τι θα κάνετε ε, για το καλοκαιρινό πακέτο και το χειμωνιάτικο πακέτο κτλ. Πρώτα απ' όλα όσον αφορά τη διακυβέρνηση, η διακυβέρνηση της, Ενεργειακής, Ενεργειακής Ένωσης. Δεν υπάρχει ακόμα σύστημα ε, διακυβέρνησης αυτής της Ενεργειακής Ένωσης, ωστόσο την προηγούμενη εβδομάδα όταν είχαμε τις συστάσεις αναχώρα ε, δεν συμπεριελήφθη τίποτα ε, για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος ενώ πέρσι σε 8 από τις ειδικέ ε, συστάσεις ε, αναφέρεται ακριβώς αυτή η φορολογική μεταστροφή, η tax shift, έτσι ώστε να βοηθηθεί η ενεργειακή πολιτική και η χρήση των ανανεώσιμων. Αλλά φέτος καμία ε, ούτε στις ε, ειδικέ συστάσεις αναχώρα, ούτε στο εξάμεινο. Καμία αναφορά ε, σε τέτοια θέματα. Υποτίθεται ότι κάθε, κάθε μέρα που περνάει βελτιώνουμε περισσότερο την κατάσταση. Αλλά και δεν καταλαβαίνω γιατί βγάζεται εντελώς τα θέματα ενέργειας και με... Ναι, ναι, αλλά αυτά θα τα δούμε αργότερα όταν θα συζητήσουμε την ε, ενεργειακή διακυβέρνηση. Όχι, νομίζω ότι από τη στιγμή που γνωρίζουμε ότι τα περιβαλλοντικά προγράμματα σχετίζονται αμεσότατα με τα, ε, τα, ε, Συγγνώμη, τα προβλήματα, τα περιβαλλοντικά συνδέονται αμεσότατα με τα οικονομικά προβλήματα, οπωσδήποτε ε... θα πρέπει να τα δούμε συνδυαστικά. Επίσης, όσον αφορά ένα από τα πέντε από τους πέντε πυλώνες στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες ε, εκπομπές ε, νομίζω ότι θα πρέπει να δείτε λίγο το θέμα της ε, μεταφοράς. Τι θα κάνετε, η ποιότητα, τι θα κάνετε με το σχιστολιθικό αέριο. Αν μιλάμε για απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές δεν είναι δυνατόν να μην το συζητάμε και αυτό. Όταν συζητάμε για το σύστημα ETS, όταν συζητάμε για εκπομπές αερίων δεν είναι δυνατόν επίσης να τα ξεχνάμε αυτά. Επίσης, αποδοτικό αποδοτικότητα, ενεργειακή αποδοτικότητα. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια όσον αφορά ε, την ε, ε, κατάσταση, γιατί ακόμα περιμένουμε τις προτάσεις όσον αφορά το τέλος των ενεργειακών καταλήπων γιατί οι αποτεφρώσεις είναι κάτι που πραγματικά θα ήταν από τα χειρότερα που θα μπορούσαν να συμβούν. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος, εξίσου σημαντικός όμως για την ομάδα EFTD. Κυρία Εύη. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας εκθέσατε ένα ιδιαίτερα φιλόδοξο πρόγραμμα όσον με, με κύριο στόχο βέβαια την μείωση της εξάρτησης από το εξωτερικό <clears throat> και την χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη. Ε, βεβαίως για να γίνουν όλα αυτά που μας λέτε θα πρέπει ε, να υπάρξουν αρκετές τροποποιήσεις, μεταρρυθμίσεις, τροποποιήσεις νομοθεσίας ας πούμε για το ETS και την ε, διαρροή και αποθήκευση η άνθρακα κτλ. Ε, το ζήτημα ε, θα ήταν να υπάρχει μια πραγματική μείωση των αερίων θερμοκηπίου <clears throat> στην ε, βιομηχανία και καταλαβαίνουμε ότι μέχρι τώρα η πολιτική έχει αποτύχει θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι εναλλακτικές στο ETS. Έχουμε επίσης και την οδηγία ε, για την ε, διαρροή και την αποθήκη και αποθήκευση του άνθρακα και εκεί προβλέπεται ε, αναθεώρηση, ρήτρα αναθεώρησης για φέτος. Αλλά μέχρι τώρα δεν έχουν δημιουργηθεί, δεν έχουν χτιστεί αυτές οι εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονται. Επίσης παραμένουν πάρα πολλά μεγάλα προβλήματα και ισχυρές αμφιβολίες για το κατά πόσο θα μπορέσει να μεταρρυθμιστεί ε, ε, το, ο τομέας αυτός. Δεν θεωρείται ότι θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξουν κάποιες νέες αποφάσεις όσον αφορά κυρίως την ε, απώλεια θέσεων εργασίας και την έλλειψη πρόδρου. Επίσης, νέες μορφές χρηματοδότησης. Δεν θα πρέπει κάτι να γίνει έτσι ώστε η χρηματοδότηση ε, να αφορά ε, την, ε, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την πλήρη τους ένταξη στο κοινοτικό ηλεκτρικό σύστημα καθώς επίσης και στη δημιουργία ευφυών δικτύων. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα τον λόγο στον Αντιπρόεδρο κύριο Σεύσκοβιτς έτσι ώστε να απαντήσει αν στις ερωτήσεις ε, που Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ όλους τους βουλευτές για τις ερωτήσεις. Τους κυρίους Λίζε Εκχάουτ που τόνισαν και τη σημασία της διακυβέρνησης και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του ρόλου του. Αναμφίβολα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλες τις νομοθετικές προτάσεις πρέπει να έχει έναν απόλυτα εξασφαλισμένο ρόλο. Αυτό είναι θεμελιώδες γιατί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι συνομοθέτης και εμείς ε, είμαστε υπόλογοι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δεν ετέθη ποτέ υπό αμφισβήτηση ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και στο πλαίσιο του συστήματος ε, διακυβέρνησης που θα ισχύσει στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για το κοινό έργο μας ε, για τις νομοθετικές προτάσεις που συνδέονται με τον τομέα της ενέργειας και την Ενεργειακή Ένωση. Θα ήθελα να επαναλάβω για μια ακόμη φορά ε, και να εξηγήσω τι σύστημα διακυβέρνηση επεξεργαζόμαστε. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι για εμάς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σημαντικό να έχουμε ένα σύστημα δυναμικό και εύρωστο, πάντα μιλάω για τη διακυβέρνηση, θέλουμε σαφείς ελέγχους, ε, παρακολούθηση, θετική ενθάρρυνση. Χωρίς αυτά δεν θα πετύχουμε ποτέ τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ταυτόχρονα όμως αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι ξεκινά κάτι καινούριο εργαζόμαστε σε ένα τομέα που για πολλά χρόνια ε, θεωρείται τομέα τομέας εθνικής κυριαρχίας παρά το γεγονός ότι ε, μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας τονίζαμε ότι εδώ μιλάμε πλέον για ε, συναρμοδιότητα και συναπόφαση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε τις προτάσεις μας. Τώρα θα υποβάλουμε τις αναλύσεις μας στα κράτη-μέλη να δούμε πώς βλέπουμε την ενεργειακή ε, νοσή και υπό το πρίσμα των κρατών μελών και τι απόδοση, τι δράσεις πρέπει να αναλάβουν, ποιες είναι οι αδυναμίες, ποια είναι τα ισχυρά σημεία για τα κράτη-μέλη, τι σημαίνει για κάθε ένα από τα κράτη-μέλη ενεργειακή ένωση. Και θέλουμε επίσης να ακούσουμε και τις δικές τους αναλύσεις, συμφωνούν με τη δική μας ε, ανάλυση, μήπως έχουν άλλες απόψεις. Υπάρχει μια κοινή βάση από την οποία μπορούμε να ξεκινήσουμε τη δουλειά μας. Και τώρα αυτή είναι η διαδικασία που έχει ξεκινήσει εντατικά και αυτό θα ισχύει από σήμερα μέχρι ότου καταλήξουμε στην υποβολή των εκθέσεων προς εμάς ε, το φθινόπορο του 2015. Φυσικά σε αυτή τη συζήτηση με τα κράτη-μέλη περιλαμβάνουμε συγκεκριμένα ερωτήματα για την ενεργειακή απόδοση, για την απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, για τους στόχους που έχουμε για το 2030 σε σχέση βέβαια και με την πορεία μας προς την εκπλήρωση των στόχων μας για το 2050, γιατί αυτό συμφωνήσαμε από κοινού. Και όλα αυτά στη συνέχεια θα τα συνθέσουμε, θα τα αναλύσουμε και θα, τα, θα, σας τα υποβάλουμε για την Ενεργή ελπίζω, του χρόνου τον Οκτώβρη. Ελπίζω να είναι ένα ενιαίο εγχείρημα, μια, μια συγγνώμη, άσκηση ένα ετήσιο εγχείρημα κάθε χρόνο να βλέπουμε δηλαδή με τα κράτη-μέλη πώς προχωρούμε, ποια είναι τα αποτελέσματα ε, με την Ευρωπαϊκή πού υπολοιπόμεθα, πού χρειάζεται περισσότερη πολιτική πίεση, ε, πολιτική όθηση. Υπουργοί ενέργειας, περιβάλλοντος, ανταγωνιστικοτητα κτλ. Ε, να τα συζητούσε στο Συμβούλιο και οι ηγέτες το Δεκέμβριο στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων και αυτοί θα δώσουν τη δική τους συνεισφορά και θα ακούσουν και το πώς, ε, τις προτάσεις για το πώς μπορούμε να προχωρήσουμε και να σημειώσουμε πρόοδο με την Ενεργειακή Ένωση. Επίσης θέλουμε να αξιοποιήσουμε και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Θεσμικών Οργάνων και των κρατών μελών στον τομέα αυτό, προκειμένου να καταλήξω σε κάτι που εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είναι φιλόδοξο, να είναι ένα εθνικό σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα. Θέλουμε να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη, να έχουμε συγκεκριμένα σχέδια, συγκεκριμένου οδικού χάρτε από τα κράτη-μέλη, για να μα πούν πώ θέλουν να πετύχουν του στόχου. Πώ μπορούν να μα βοηθήσουν επίση να οικοδομήσουμε ε, από την Εθνική Σκοπιά την Ενεργειακή Ένωση. Αυτό είναι λοιπόν το σχέδιο, αυτή είναι η πρόθεσή μα. θα υποβληθούν συστάσεις σχέση με αυτά τα εθνικά σχέδια για το κλίμα και την ενέργεια και σε αυτά θέλουμε να περιληφθούν συστάσεις οι οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται στις συστάσεις αναχώρα στο πλαίσιο των μακροοικονομικών, της μακροοικονομικής δέσμης μέτρων για φέτος. Θέλουμε λοιπόν οι συστάσεις αναχώρα να ε, εστιάσουν στην απασχόληση, τα μακροοικονομικά ζητήματα και όλα τα σχετικά ζητήματα που είναι πιο εξορθολογισμένα για τα κράτη-μέλη. Αλλά δεν λησμονούμε ότι σε ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις που αναφέρατε, σε πολλέ περιπτώσει, σε πολλά κράτη-μέλη υπάρχουν διευθυντές γραμμέ για τι κρατικέ ενισχύσει, για την ενέργεια ιδίω. Για τη σταδιακή κατάργηση των επιβλαβών για το περιβάλλον επιδοτήσεων. Και όλα αυτά τα μελετούμε και θα τα επεξεργαστούμε στι μελλοντικές μα συστάσεις σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη για τα εθνικά σχέδια και τα ενεργειακά σχέδια. Έρχομαι στον δόκτωρα Λίζε γιατί θα ήθελα να συμπληρώσω τις πληροφορίες για αυτό το νέο σύστημα διακυβέρνησης και το πώς σχετίζεται αυτό με την κατάσταση της Ενεργειακής Ένωσης και τα εθνικά σχέδια δράσης για το κλίμα και την ενέργεια. Σε ό,τι αφορά την ενεργειακή απόδοση φυσικά και θα επεξεργαστούμε την αναθεώρηση της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση έχοντας υπόψη μας το στόχο του 30% όπως αυτό το υπογράμμισε και το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα συμπεράσματά του. Αυτή είναι η πρότασή μας και πιστεύει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι αυτή είναι η σωστή οδός. Δεν θέλουμε να μας διαφύγει το γεγονός ότι ακόμη και το 25% το έχει θεωρήσει το Ευρωπαϊκό Συμβουλίο σαν πρωτογενή στόχο. Είναι σαφής λοιπόν ε, η φιλοδοξία μας και ελπίζω η συμφωνία στο Παρίσι να ανοίξει το δρόμο και για μια πιο φιλόδοξη προσέγγιση. Τι πρέπει να περιμένουμε από το Παρίσι τώρα. Πιστεύω ότι θα μιλάμε για επιτυχία στο Παρίσι αν έχουμε μια συμφωνία που θα είναι νομικώς δεσμευτική κατά προτίμηση δε θα έχει μία μορφή πρωτοκόλου UNFCC, ένα πρωτόκολλο που έπειτα θα πρέπει να τεθεί σε ισχύ το συντομότερο δυνατό εφόσον το επικυρώσουν οι χώρες που το 80% των εκπομπών ε, το 2010 και υπάρχει και μια δυναμική θέλουμε να υπάρχει τακτική αναθεώρηση και επανεξέταση ε, τηρούμε τους στόχους, μειώνουμε ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα συνολικά παίρνουμε τα ε, σωστά μέτρα, είναι, τηρείται το χρονοδιάγραμμα υπάρχει επαρκή της διαφάνεια δίνουμε, ε, έχουμε αποτελέσματα τα οποία είναι Εντό των προθεσμών που έχουμε θέσει. Αυτά όλα θα κρίνουν την επιτυχία. Στο Παρίσι, αν συμφωνηθούν αυτά δηλαδή. Ελπίζουμε βέβαια ότι όλο και περισσότερες χώρες ε, θα κάνουν αντίστοιχες προτάσεις. Εμείς τους στόχους μας τους παρουσιάσαμε και ελπίζουμε και πολλές άλλες χώρες να ακολουθήσουν τα βήματά μας από τις χώρες εννοώ που συμμετέχουν σε αυτές τις ε, διαπραγματεύσεις σε ό,τι αφορά τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς που θα υποβάλουν. Έχουμε και τους ε, σημαντικούς ε, φορείς εκπομπών, θα συνεργαστούμε με τις σημαντικότερες χώρες για να δημιουργήσουμε πρόσφορο έδαφος για μια συμφωνία στο Παρίσι. Βασικός διαπραγματευτής είναι ο Μιγέλ Αρεσκανιέτε που σημαίνει στο Βερολίνο για συνομιλίες θα συμμετάσχει στο G7, στο G7 αύριο στην υπορκή διάσκεψη στο 7 και με βέβαιος ότι θα ηγηθεί και με τον καλύτερο τρόπο τη διαπραγματευτική μα ομάδα στο Παρίσι. Τώρα, κατά τα λοιπά, εμεί στην οικογένεια τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια. Έχουμε ε, σχεδιάσει διπλωματική διπλωματικές πρωτοβουλίες για να προσεγγίσουμε τα κράτη της πόλης. Έχουμε το πρόγραμμα των εφιών πόλεων. Θέλω να δραστηριοποιηθώ και εγώ και όλοι θα κάνουμε πάντα δυνατόν ώστε όλοι ε, να συνεισφέρουμε προς ε, την επιτυχία της διάσκεψης του Δεκεμβρίου στο Παρίσι. Σε ό,τι αφορά το ETS, την εμπορία εκπομπών, φέτος το καλοκαίρι, να σας πω κύριε Γκρότε, και μάλιστα πριν ε, διακόψουμε για τις θερινές διακοπές, θα έχουμε κάποιες εξελίξεις, θα κοιτάξω πολύ κοντά και τα θέματα της διαρροής άρθρακα. Είναι πολύ σημαντικό για το Κοινοβούλιο, για σε ό,τι αφορά την ε, αποτροπή αυτής της ε, διαρροής, να υπάρχει σχετική πρόβλεψη, αλλά θα πρέπει να μπει και στο σωστό πλαίσιο για να αντικατοπτρίζονται τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και δυνατότητες τα τελευταία πιο πρόσφατα κριτήρια τα οποία έχουμε υιοθετήσει ώστε το σύστημα ETS θέλουμε να είναι και φιλόδοξο αλλά και να μην οδηγεί σε διαρροή άνθρακα από την Ευρώπη σε άλλες χώρες και σε ό,τι αφορά τα διελιστήρια. Είναι πολύ σημαντικό να υπογραμμίσουμε ότι για τον κλάδο αυτό είχε σημαντικό να γίνουν αποδεκτέ κάποια, κάποια κριτήρια και όρια αναφοράς ε, πολύ σημαντικά. Αυτή η προσέγγιση είναι σημαντική και στο πλαίσιο αυτών των μεταρρυθμίσεων του ETS. Ε, θα εξετάσουμε και τον δεχόμενο διαφοροποιήσεων. Θα δούμε και την έκθεση των βιομηχανιών ε, σε πιθανό ανταγωνισμό από χώρε και εδάφη όπου δεν υπάρχει τόσο απαιτητική νομοθεσία. Έρχομαι στον κύριο Γκερμπράντι για την ανταγωνιστικότητα. Συμφωνώ μαζί σας ότι είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα η Ευρώπη της αποσύνδεσης της οικονομικής ανάπτυξης και της μείωσης, από τη μείωση μάλλον των εκπομπών. Είχαμε το στόχο να μειώσουμε από το 90 και μετά τις εκπομπές ε, το πετύχαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό και αυτό δείχνει τη δική μας θετική εμπειρία ότι δηλαδή όταν μιλάμε για ενεργειακή απόδοση εταιριών εδώ έχουμε διπλάσια απόδοση σε σχέση με τις ε, βιομηχανίες ε, των ΙΠΑ και αυτό είναι σημαντική συνεισφορά για το μέλλον για τη συνολική αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα των εταιριών μας. Και νομίζω ότι αυτό το αντιλαμβάνονται όλο και περισσότερο τα κράτη-μέλη. Για να τα πείσουμε στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης να ακολουθήσουν αυτή την ε, αντίληψη και να θετήσουν μια ευρωπαϊκή προσέγγιση δεν θα είναι εύκολο βέβαια. Όμως πρέπει να εστιάσουμε στην, στο επιχείρημα ότι μπορεί η, Ευρωπαϊκή, η Ενεργειακή Ένωση να είναι μια διαφορετική πρόπτικη για τις βόρειες σκανδιναβικές χώρες για παράδειγμα να αφορά πιο πολύ ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ενεργειακή απόδοση, ενώ για τις νοτιοανατολικές ευρωπαϊκές χώρες να αφορά περισσότερο την ε, ενεργειακή ασφάλεια, για τις χώρες κεντρικής Ευρώπης, την περιφερειακή συνεργασία και το καθεξής. Κάθε χώρα θα εστιάσει κάπου διαφορετικά ενδεχομένω. Όμως, ταυτόχρονα θα πρέπει να φροντίσουμε αυτές τις διαφορετικές προπιές να τις ε, ε, βάλουμε κάτω από την ίδια ομπρέλα, κάτω από μια κοινή πολιτική. Οι ιδιαιτερότητες των χωρών να οδηγήσουν σε μια πιο αποδοτική προσέγγιση και μέτρα και αποτελέσματα θετικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Τάμιο Επενδύσεων Juncker. Ξέρω ότι πολύ σύντομα θα έχουμε ένα τριμερή διάλογο για το θέμα αυτό και ο συνάδελφος Κατάινεν και η συνάδελφος Γεωργίευα θα συμμετάσχουν. Ελπίζω να επιτευχθεί σημαντική πρόοδο σε αυτόν τον τριμερή διάλογο. Τώρα, για τα έργα του μέλλοντος, αυτό που λείπει στην Ευρώπη εκεί που δεν είναι επαρκής οι επενδύσεις είναι οι ε, υποδομές ε, στον τομέα της ενέργειας και των μεταφορών. Γνωρίζω ότι είναι πολύ σημαντική για την Επιτροπή σας ενεργειακή απόδοση και για το Κοινοβούλιο εν γέννη. Είμαι βέβαιος ότι η ενεργειακή απόδοση θα είναι ένα σημαντικό τομέας όπου μπορεί να έχουμε επενδύσεις σημαντικές ε, προερχόμενες από το Ταμείο Επενδύσεων του Γιούνκερ και στο τέλος είμαι βέβαιος ότι θα εξασφαλιστεί αυτή η χρηματοοικονομική υποστήριξη, θα είναι εξισορροπημένη βέβαια μεταξύ όλων των προτεραιοτήτων που πρέπει να λάβουμε υπόψη στην τρέχουσα περίοδο. Και τώρα, μου επιτρέπετε, να καταλήξω πατώντας τα επόμενα ερωτήματα για την κυρία Κονέτσνα. Νομίζω απάντησα ήδη για τη διαφοροποίηση δηλαδή των ενεργειακών ε, πηγών. Εργαζόμαστε σκληρά, ώστε οι παραδοσιακέ ενεργέ πηγέ που έχουμε από Ρωσία, Νορβηγία, Αλγερία, να συνδυαστούν να με το διάδρομο και το διάδρομο της Κασπίας και βέβαια και για το υγραέριο. Θέλουμε και αυτό να συνεισφέρει για να συμπληρώσει τους ενεργικούς ε, πόρους, ενεργικές πηγές και βέβαια και η ενεργειακή απόδοση, είναι σημαντική ως αρχή. Στην αρχή δηλαδή σε, κάποιο, οποιοδήποτε project πρέπει να μετρήσουμε τη δυναμικότητα, τη χωρητικότητα, να κάνουμε προβολές για το 2020, 2025, 30, τα ορυκτά καύσιμα ε, κτλ. Και να αξιολογήσουμε τις ανάγκες για πρόσθετες υποδομές ενδεχομένως. Η ενεργειακή παινία, ενεργειακή φτώχεια είναι κάτι πολύ σημαντικό και θα συνεργαστούμε στενά με τα κράτη-μέλη για να αντιμετωπίσουμε με το καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόβλημα. Θέλουμε το πρόβλημα της ενεργειακής παινίας να το αντιμετωπίσουμε ίσως ε, με τις ε, τιμές της ενέργειας, με την τιμολόγηση ή με κάποια συγκεκριμένα προγράμματα στα κράτη-μέλη που έχουν πρόβλημα περισσότερο. Να υπάρχει ίσως ένα κοινωνικό τιμολόγιο ή ένα είδος υποστήριξης για όσους χρειάζονται βοήθεια. Χωρίς αυτό να οδηγήσει βέβαια σε στρέβλωση της εσωτερικής αγοράς. Στον κύριο Eichhout τώρα και στην κυρία Εύη να πω ότι η απαλλαγή ε, των ε, μεταφορών από τις ε, εκπομπές άνθρωποι για το 2016-2017 είναι ένα θέμα με το, για το οποίο εργαζόμαστε στην με, με τον κύριο Μπούλ και αυτά τα, τις μονάδες επίδειξης είναι μια τεράστια επένδυση, κοστίζει πολλά χρήματα. Είναι προτεραιότητα στον τομέα της έρευνας, στην ενέργεια. Στον Καναδά μόνο έχουμε δει ένα επιτυχημένο παράδειγμα μέχρι τώρα, αλλά έχω δει πρόοδο και στην Ευρώπη σε ορισμένα σχετικά project και πρέπει να τα ενθαρρύνουμε και να δούμε και πώς μπορούμε να τα χρηματοδοτήσουμε με τα νέα αυτά ταμεία. Δεν ξέρω αν έχω παραλείψει κάποια ερωτήματα. Προσπάθησα να απαντήσω σε όσο το περισσότερο ερωτήματα των συντονιστών. Εμείς σας ευχαριστούμε για την απάντησή σας. Τώρα θα ζητήσω από τους συναδέλφους που θα πάρουν το λόγο να μην ξεπερνούν το 1,5 λεπτό που έχουν στη διάθεσή τους και θα δώσω αμέσως το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Merci beaucoup. Σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, όντως μας έχετε δώσει ήδη πολλές πληροφορίες. Ε, για ένα θέμα πολύ σημαντικό που αφορά την ε, Ενεργειακή Ένωση. Αναφερθήκατε στην διαφοροποίηση, αναφερθήκατε στο σχέδιο της ε, μεταφοράς του, της ενέργειας από την Κασπία, αλλά εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, δεν μιλάτε καθόλου για την Μεσόγειο. Είναι μια πολύ πλούσια ε, περιοχή και όσον αφορά τις ενεργειακές ε, ευκαιρίες, ανανεώσιμες πηγές όπως είναι ο, ο, ε, ήλιος, αλλά και η ηλιακή ενέργεια, αλλά και όπως είναι οι δυνατότητες μεταφοράς μέσω της Μεσογείου. Δεν θα έπρεπε να ξεκινήσει κάποια συνεργασία και με την Μεσόγειο και με τις χώρες της Βόρειας Αφρικής, χώρες Μαχρέμπ, έτσι ώστε να ενδυναμωθεί αυτή η έννοια της διαφοροποίησης. Ευχαριστώ πολύ η κυρία Ντάλι. Thank you, Chair. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, μας είπατε σήμερα και σας ακούσαμε με προσοχή να μας λέτε και να μας αποδεικνύετε ότι υπάρχει ισχυρή βούληση από πλευρά της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έτσι ώστε να στεφθεί από επιτυχία η Ενεργειακή Ένωση. Εγώ αναφέρομαι τώρα στην δέσμη και ε, της ε, Ενεργειακής Ένωσης ε, και για πρώτη φορά γίνεται σε αυτή λόγος για την απαλλαγή <clears throat> από την ε, ε, τις ανθρακούχες εκπομπές. Ε, αναφέρονται ήδη τα θέματα αυτά στα συμπεράσματα του Ενεργειακού Συμβουλίου του Μαρτίου, πράγμα πολύ σημαντικό. παρόλα αυτά θα πρέπει να εισαχθούν όσο γίνεται γρηγορότερα κάποια νομοθετήματα όσον αφορά την ασφάλεια του ανεφοδιασμού, όσον αφορά τις διευρυμένες δυνατότητες αποθήκευσης αλλά και την αλληλεγγύη πόσο πολύ θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιτύχει ε, αυτούς τους στόχους ε, της αηφορίας ε, και της απαλλαγής από τον άνθρακα ε, ε, νομίζω ότι θα πρέπει να προτείνεται και, ε, και ναι, κάποιο εναλλακτικό οδικό χάρτη όσον αφορά την μεταφορά ενέργειας, όσον αφορά και την χρήση εναλλακτικών μορφών ενέργειας για την δημιουργία ηλεκτρισμού που θα είναι σημαντικό για το μέλλον. Ευχαριστώ πολύ. Ντάνκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Πρέπει να έρθετε στη σκοτία κάποια στιγμή γιατί η Ενεργειακή Ένωση ε, λειτουργεί εκεί σε μικρή κλίμακα δηλαδή σε ό,τι αφορά διασυνδέσεις ε, ανανεώσιμες κλπ. Τώρα για την ε, Κανονική Ενεργειακή Ένωση ε, μου θυμίζει τους τυφλούς που ακουμπάνε ένα κομμάτι του ελέφαντο καθένας και περιγράφουν διαφορετικά πράγματα. Δηλαδή, άμα πάμε να μιλήσουμε σε κάποιο κράτος μέλος, μετά σε άλλο, θα δούμε κάτι παρόμοιο να συμβαίνει. Τώρα μας τραβάει σε μια κοινή θέση η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά δεν υπάρχει κοινότητα στόχων και θέσεων. Διατρέχουμε κίνδυνο να φτιάξουμε 28 διαφορετικές διακριτές ενεργειακές ενώσεις εγώ νομίζω ότι το δίκτυο της Βόρειας Θάλασσας ε, ε, θα πρέπει να το δούμε καλύτερα γιατί είναι ένα καλό παράδειγμα ε, για το πώς μοιράζουμε την ενέργεια, πώς την επιμερίζομαι. Θα πρέπει όμως να προσεγγίσουν πρώτα κάποιους κοινούς στόχους το, τα κράτη-μέλη και να βρεθεί και μία προσέγγιση χρηματοδοτική ρεαλιστική γιατί αν δεν, ανα, δεν τέτοιου είδους δεσμεύσεις ε, θα μείνουμε στην κατάσταση των ανθρώπων που ο καθένας πιάνει και συνειδητοποιεί διαφορετικό κομμάτι του ελέφαντα. Η κυρία Τόγκρες Μαρτίνες. Ευχαριστώ πολύ. Τα ωφέλη του συστήματος διαχείρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα εφαρμοστεί είναι αμφίβολα για τους πολίτες η στρατηγική για την ενέργεια που προωθεί η Κομισιόν με τη δημιουργία ενιαίας ε, αγοράς ενέργειας και ενίσχυων διασυνέσεων μεταξύ τα κράτη βασίζεται σε ένα σύστημα με μεγάλα κέντρα παραγωγής και μεγάλα κέντρα κατανάλωσης, αλλά βασίζεται σε φυσικό αέριο που δεν έχουμε. Βάσει τους υπολογισμούς αυτό το σχέδιο απαιτεί 200 δις ευρώ επενδύσεων για την επόμενη δεκαετία για να φτάσουμε στο 10% το πολύ διασύνδεση μεταξύ των κρατών με την κατά κατασκευή αγωγών και γραμμών υψηλής τάσης. Πώς αυτά τα σχέδια υποδομών μπορούν να ωφελήσουν τις επιχειρήσεις και τις οικογένειες, πολλές εκ των οποίων βλέπουν ότι οι δυνατότητες επενδύσεων και η αγοραστική τους δύναμη μειώνονται λόγω ε, καταχρηστικό πρακτικό στον τομέα της τιμολόγησης. 51 ε, εκατομμύρια πολίτες σύμφωνα με στοιχεία της Γιώργης δεν πληρώνουν το ρεύμα, δεν μπορούν να το πληρώσουν. Και τελικά θα οδηγηθούμε με αυτή την Ενεργειακή Ένωση σε κοινωνικό αποκλεισμό. Εμείς δεν μπορούμε ως πολιτικοί να το ανεχθούμε. Γι' αυτό λοιπόν ε, είναι σαφό, σαφό, σαφές ότι εμείς έχουμε επιφυλάξει για αυτό το μοντέλο και σας ζητούμε να επαναπροσανατολίσετε αυτές τις προτάσεις σε ένα μοντέλο που θα βασίζεται στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και ανάπλαση του περιβάλλοντος, του αστικού και των ε, ε, μεταφορών, ε, να στηρίξετε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, δημοκρατική διαχείριση, ισορροπία μεταξύ των δικτύων και καθολική πρόσβαση στην ενέργεια. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Αντιπρόεδρε. Επανέρχομαι στο θέμα της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές που είναι πολύ σημαντικό κομμάτι, το πιο σημαντικό στην Ενεργειακή Ένωση. Είναι... Οι επιδοτήσεις όμως που είναι ζημιογόνες πολλές φορές και δεν συμβάλλουν στην εξάλληψη του άνθρακα γίνεται μία ε, καυτή συζήτηση για την ενεργειακή ασφάλεια που είναι απόλυτα δικαιολογημένη βέβαια αφού τα κράτη-μέλη θέλουν ε, ασφάλεια στην ενέργεια. Αυτή η συζήτηση όμως άλλες φορές χρησιμοποιείται ως δούριος ύπος ε, υπέρ της γηγενούς παραγωγής βλέπε σχή στο λιθικό αέριο για παραγωγή ενέργειας, ε, για θέρμανση ψήξη και άλλα ορυκτά καύσιμα επίσης. Ερωτώ λοιπόν πώς θα εναρμονίσετε τις ανάγκες των κρατών μελών στον τομέα της ασφάλειας της ενέργειας με στόχο μια απαλλαγή από ανθρακούχες εκπομπές όταν καμιά φορά στη, και στην κεντρική και ανατολική Ευρώπη και νοτιοανατολική τα θέματα ενεργειακής ασφάλειας φαίνεται ότι υπερισχύουν του θέματος της βιωσιμότητας και της απαλλαγής από ανθρακούχες εκπομπές. Οι προτεραιότητες δηλαδή μπαίνουν διαφορετικά. Ευχαριστώ κύριος Φόντε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι λύσεις οι οποίες ε, αφορούν ε, την ενεργειακή ασφάλεια θα πρέπει ε, να ολοκληρωθούν λαμβάνοντας υπόψη όλες τις ανάγκες με ισορροπημένο τρόπο. Ε, καλοδεχούμενες είναι οι προτάσεις της Κομισιόν που φαίνεται ότι βάζουν στο κέντρο τους, έχουν στο κέντρο τους τον πολίτη, πράγμα που μας ευχαριστεί. Όσον αφορά τους πολίτες θα έχω λιγότερο τεχνικής φύσεως ε, ερωτήσεις ε, γιατί εγώ ζήτησα τους πολίτες να μου πούν τι θα σας ρωτούσαν αν σας είχαν μπροστά του. Επομένως σας ρωτώ, προβληματίζονται οι πολίτες για από την από την ε, από την ενεργειακή εξάρτηση από την Ρωσία και την Αφρική. Δεύτερη ε, ερώτηση, ανεξάρτητοι ερευνητές, ε, ανεξάρτητοι εννοώ από τις πετρελαϊκές ε, εταιρείες, προβλέπουν ότι θα υπάρξει μία κορύφωση της χρήσης του πετρελαίου τα επόμενα χρόνια. Έχετε μία άποψη και κάποια στρατηγική όσον αφορά το θέμα αυτό. Τρίτον, ξέρουμε ότι ε, δεν πέρασε στην Ήτρε η τροποποίηση όσον αφορά την ε, υδρορογμάτωση, ε, το fracking και επομένως έχετε κάποια άποψη όσον αφορά την χρήση αυτής της υδρορογμάτωσης του fracking στην τόσο πυκνοκατοικημένη Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Σπέντερλετ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, η παρουσίασή σας ε, μου ανέβασε τα επίπεδα ενέργεια σήμερα. Προτείνω στην Κομισιόν μαζί με τα κράτη-μέλη να αρχίσουν να αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο επενδύουμε δημόσιο χρήμα στην ανάπτυξη της υπαίθρου και να το δει ως κομμάτι της ενεργειακής ε, ε, Ευρώπης γιατί οι μικροί αγρότες έχουν μικρά εισοδήματα, λίγο κέρδος και υψηλό κόστος ενέργειας. Στη Σλοβενία να σας εξηγήσω. Επενδύω και επιδοτούμε ε, για την παραγωγικότητα ε, της γεωργίας χωρίς όμως να αλλάζουμε την ενεργειακή διάρθρωση. Πώς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι επιδοτήσεις λοιπόν, δεν πρέπει να δώσουμε κίνητρα για να επενδύσουν οι γεωργοί, οι αγρότες στις ε, ανανεώσιμες ε, θα πρέπει να γίνει με ε, έξυπνο τρόπο. Με εγγυημένες τιμές μπορεί να βάλει συστήματα ηλιακής ενέργειας και να, έχει, να λάβει δάνεια με ευνοϊκούς όρους. Εν τω μεταξύ θα προσαρμόζονται ε, στις, ε, στα νέα μηχανήματα. Οι επιδοτήσεις θα δίνονται απευθείας στην παραγωγή ενέργειας. Αυτό μπορεί να γίνει. Τέλος, ε, μια τέτοια ενέργεια που θα λαμβάνει υπόψη και το κλίμα θα πρέπει να ενταχθεί σε μια νέα στρατηγική σε επίπεδο ένωσης. Έτσι το αντιλαμβάνομαι. Κύριε Αντιπρόεδρε, μπορεί να γίνει τα επόμενα χρόνια μια τέτοια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκούτελάντε. Ευχαριστώ. Ε, πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε για την εξαιρετική παρουσίαση με πολλά στοιχεία και ε, ευχαριστώ και για τη σαφήνεια στις απαντήσεις σας μετά τον πρώτο γύρο ερωτήσεων. Χαίρομαι που μιλήσατε για την ανανεώσιμη ενέργεια και θέλετε και μια οδηγία το 2017 ή το 2018. Για, υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι για τη στρατηγική 2030 για τις ανανεώσιμες, αλλά στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Οκτωβρίου ένα νέο μοντέλο αναφέρεται που θα έχει σε επίπεδο νοσιακό δεσμευτικούς στόχους ένα νέο μοντέλο ελέγχου της ε, εφαρμογής αυτών των μέτρων. Όμως πώς θα συνεχιστεί η προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να ξεπεράσουμε τους πρώτους στόχους και πώς θα φροντίσουμε και άλλοι μηχανισμοί να στηρίζουν το έργο της Ένωσης στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας όπως ας πούμε το πρόγραμμα επενδύσεων για τους ε, νέους αγρότες. Πώς μπορεί όλοι αυτοί οι τομείς να συμβάλλουν σε αυξανόμενη χρήση ανανεώσιμων γιατί δίνουμε έμφαση στην ασφάλεια του εφοδιασμού ενώ πρέπει να συμπεριλάβουμε τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην οικοδόμηση της Ενεργειακής Ένωσης. Ευχαριστώ, κυρία Σουίτσα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, κυρία Αντιπρόεδρε. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την αρχική παρουσίαση που ήταν σαφέστατη, πολύ καλά δομημένη και εύκολη είναι η συναγωγή των συμπερασμάτων. Βέβαια η εισαγωγή σας ήταν αρκετά γενική και όλοι γνωρίζουμε ότι η Ενεργειακή Ένωση είναι ένα εγχείρημα πολύ φιλόδοξο με στόχο την εναρμόνιση του εφοδιασμού σε ενέργεια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρατε και διάφορους τρόπους για την επίτευξη των στόχων, διάφορες διαστάσεις, τη σκέλη, το πολιτικό, την πολιτική διάσταση, την διπλωματική, την νομοθετική διάσταση. Για την πολιτική διάσταση, αναφέρατε την, ε, το δημόσιο διάλογο που θα γίνει στα κράτη-μέλη, ώστε να συμπεριληφθούν όχι μόνο οι τοπικοί εμπλεκόμενοι, βαθμό όπως οι δήμαρχοι αλλά και μη κυβερνητικέ οργανώσεις και άλλοι εμπλεκόμενοι που πρέπει και αυτοί να συμμετέχουν ενεργά στο εγχείρημα της Ενεργειακής Ένωσης. Ερώτηση λοιπόν, πώς σχεδιάζετε να λύσετε το ακόλουθο πρόβλημα. Οι εφοδιαστές ενέργειας ελέγχουν στην ουσία τις τιμές της ενέργειας. Και κυριαρχούν με την έννοια ότι είναι και ιδιοκτήτες πολλών πηγών ενέργειας. Δεύτερη ερώτηση. Ε, η χρήση της ενέργειας. Έχουμε δεσμευτικούς... Ε, α, τα ορυκτά καύσιμα. Έχουμε δεσμευτικούς στόχους, ε, αλλά ε, πώς θα ε, εκπληρώσουμε, πώς θα πραγματοποιήσουμε αυτούς τους στόχους, τους δεσμευτικούς. Ε, τώρα, ε, εγώ είμαι από την Κροατία. Πότε στην Νοτιοανατολική Ευρώπη θα πάρουν οι πολίτες συγκεκριμένες πληροφορίες για τον Αδριατικ, το βραχίωνα της Αδριατικής ε, αυτού του αγωγού. Γιατί μέχρι τώρα εμείς δεν έχουμε ενεργειακή ασφάλεια στον εφοδιασμό. Ε, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πρόοδες που έγιναν για το πρόγραμμα τερματικού του υγραερίου που είναι, έχει συμπεριληφθεί στο πρόγραμμα Juncker. Τι προβλέπετε εδώ, πότε θα αρχίσει το έργο να υλοποιείται, δηλαδή η καθ' αυτό κατασκευή πότε θα αρχίσει, γιατί περιμένουμε αυτό το, το σχέδιο, το έργο, ότι θα είναι ευκαιρία δημιουργίας θέσεων εργασίας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να σας ρωτήσω την, ε, να μου πείτε τη θέση σας όσον αφορά την συνεχιζόμενη χρήση των ε, ορεικτών καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι ξέρουμε ποιες είναι οι σκέψεις ε, για το κλίμα, όλοι μας γνωρίζουμε ότι υπάρχουν κάποιες επιπτώσεις, ε, αλλά τα ορυκτά καύσιμα, κυρίως δε ο άνθρακας, συμμετέχουν, ε, με, συμμετέχουν με πολύ σημαντική θέση ε, στο ενεργειακό μείγμα ορισμένων χωρών. Δεν γίνεται να αλλάξει μέσα σε μία μέρα η κατάσταση αυτή αλλά η, ε, και επιπτώσεις μια γρήγορης ε, τροποποίησης μπορεί να είναι μεγάλες. Η γρήγορη λοιπόν μετακίνηση προς ένα άλλο ε, τρόπο ενέργειας που δεν θα έχει τόσες πολλές εκπομπές σε μια πρώτη φάση οπωσδήποτε θα σημάνει ε, αύξηση της ε, εισαγωγής αερίου και θα υπάρχουν προβλήματα όσον αφορά τις πρώτες ύλες και την εισαγωγή τους και σε σχέση και με το θέμα της Ρωσίας. Αναφερθήκατε στην διαφοροποίηση των τιμών ενέργειας. Ε, το, η δυνατότητα αναθεώρησης του κύριου παρόχου εξανατολών που είναι η Gazprom μπορεί να ε, δημιουργήσει έτσι μια διαφοροποιημένη ε, τιμολογιακή πολιτική αλλά βεβαίως γνωρίζουμε ότι υπάρχει κάποια διαφωνία μεταξύ Gazprom και Ευρωπαϊκής Επιτροπής όσον αφορά τα θέματα αυτά. Μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω παραπάνω για τη διαφωνία με την Κάστρο. Με ευχαριστώ πολύ ο κύριος Μπέλετ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την σαφή σας παρουσίαση. Θα επανέλθω στη μεταρρύθμιση του συστήματος εκπομπών ε, ε, Αναλλαγής και εμπορίας εκπομπών ETS. Το πρώτο βήμα ήταν ε, καλό, επιτυχές και βεβαίως περιμένουμε και τα επόμενα φιλόδοξα βήματα και όσον αφορά βέβαια και το σύστημα CCS διαρροής και αποθήκευσης ε, ε, άνθρακα δύο συγκεκριμένες ερωτήσεις ε, όσον αφορά τα, τις προσόδους από το ETS. Είναι ένα ευαίσθητο θέμα ε, είναι πιθανό να ε, προκύψει ένα σύστημα κινήτρων έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να πάρουν ε, τα, τις προσόδους αυτές, τα, τα κονδύλια αυτά και να τα επενδύσουν σε κοινά προγράμματα περιβαλλοντικά. Αυτό θα ήταν μια καλή ιδέα. Όσον αφορά δε το εύρος του ETS, ε, του συστήματος εμπορίας, ε, κυρίως αφορούν οι προτάσεις ε, της μεταφορές, των τομέα των μεταφορών. Πώς βλέπετε αυτές τις προτάσεις τροποποίησης. Πρόεδρος, νομίζω ότι έχω τώρα τον κύριο Μάτσο που έχει ζητήσει τελευταίο το λόγο. Thank you, Chair. Um, Ευχαριστώ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα καταρχάς να συγχαρώ τον Αντιπρόεδρο. Σίγουρα δεν είναι το πιο εύκολο χαρτοφυλάκι αυτό που έχει αναλάβει, το διαχειρίζεται πάντως ε, άριστα με χάρη και γοητεία. Θα ήθελα να τον ρωτήσω, εξ όσων γνωρίζω, οι κοινέ δέσμες ε, ενεργειακών που θα πρέπει να είναι κάτι θελοντικό για τα κράτη-μέλη. Δεν ξέρω αν αληθεύει αυτό και τι μεχανισμοί θα ισχύσουν. Θα υπάρξει ένα πλαίσιο, μια πλατφόρμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπου θα συζητούνται τα διάφορα συμφέροντα. Και ένα άλλο ερώτημα, πώς πιστεύετε ότι θα κρατήσουμε στο τον πιο χαμηλά τις τιμές της ενέργειας σε σύγκριση ή μάλλον σε σχέση με την ανταγωνιστικότητα. Και τώρα έρχομαι στην μες πηγές ενέργειας. Πώς μπορούμε να δώσουμε κίνητρα στον κλάδο αυτό. Προβλέπετε στήριξη σχεδιασμένη για αυτό το τομέα ή θα εστιάσετε κύριο στην ενεργειακή απόδοση και τα σχετικά. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιπρόεδρε, έχετε τώρα το λόγο. Για να δώσετε πολλές απαντήσεις πάλι. Καλή τύχη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Εκτιμώ ιδιαίτερο το ενδιαφέρον και τις πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις, γιατί πολλές φορές όταν κανείς ακούει ένα ερώτημα, αντιλαμβάνεται ότι δεν έχει όλες τις απαντήσεις, ότι πρέπει να επεκταθεί πολύ. Άλλωστε βέβαια αυτός είναι και ο στόχος ε, του διαλόγου που έχουμε μαζί, να προωθήσουμε δηλαδή τις κοινέ μας πολιτικές και είμαι ευγνώμων στους βουλευτές γι' αυτό. Να απαντήσω στην κυρία Γκροστέτ. Στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις αναφέρθηκα θα έλεγα, ε, στις πρόσφατες διπλωματικές προσπάθειες που καταβάλαμε μαζί με τον ε, Επίτροπο Κανιέτε, ο οποίος επισκέφθηκε τη Λεκάνη της Μεσογείου, διάφορες χώρες της περιοχής επισκέφθηκε, σε συνέχεια της Μεσογειακής Πλατφόρμας που δημιουργήσαμε με όλες τις χώρες της λεκάνης της Μεσογείου για να ε, δούμε τα θέματα της ενεργικής ασφάλειας, ε, των διασυνδέσεων ε, για το ηλεκτρικό ρεύμα και για την αξιοποίηση του δυναμικού την ανώσουμε πηγών ενέργειας σε την περιοχή αυτή και νομίζω ότι αυτή η επίσκεψη στέφθηκε με επιτυχία. δόθηκαν σαφή ξεκάθαρα μηνύματα και από την Αλγερία και από άλλες χώρες περιοχής που είπαν ότι θέλουν να συνεργαστούν μαζί μας στα συγκεκριμένα αυτά έργα και σχέδια και είπατε και εσείς ότι υπάρχουν δυνατότητες ε, για τις ανανέσιμες πηγές ενέργειας, ιδίως ε, αιωλική ενέργεια, αιωλικές τεχνολογίες, συγγνώμη, ηλιακές ε, τεχνολογίες στην περιοχή αυτή και σίγουρα η Μεσόγειος παραμένει μία από τις περιοχές κλειδιά όπου θα αναστήσουμε ενεργειακή συνεργασία για το μέλλον. κυρία Ντάλη Μίλησε για την ε, απαλλαγή από τις εκπομπές άνθρακα, δεν ήταν ε, το μόνο θέμα, γιατί μίλησε και για τις μεταφορές και νομίζω ότι και άλλα βουλευτές απασχολεί το ίδιο θέμα. Να κάνω λοιπόν κάποια σύντομα σχόλια, γιατί σίγουρα είναι τεράστιο αυτό το θέμα και ο αρμόδιος ε, για τις μεταφορές επίτροπος είναι άκρος απασχολημένος βέβαια με όλα αυτά. Συνεργαζόμαστε πάντως και για την ανάπτυξη ε, των σταθμών για αναλεκτικά καύσιμα. Επίσης, στην αιρεσιμότητα, σε ό,τι αφορά δηλαδή, τις μελλοντικές υποδομές και τα σχετικά έργα, ιδίως για οδικές μεταφορές, περιλαμβάνουμε την ηλεκτροδότηση. Λέμε ότι θα πρέπει να εντάσσεται στις υποδομές, πρέπει να ξεπεράσουμε τα σημερινά προβλήματα. Εγώ δεν μπορώ να αγοράσω ένα ηλεκτρικό όχημα γιατί δεν μπορώ να το φορτίσω. Οι άλλες εταιρείες λένε ότι δεν θα δημιουργήσουν αυτούς τους σταθμούς φόρτισης γιατί δεν υπάρχουν αρκετά ηλεκτροκοχήματα Προς και πίσω ρέμα. Και πρέπει να υπάρξει πρόοδος και να είναι συνεχή, σταθερή, να ρέει και αν πραγματικά χρησιμοποιούμε την ευρωπαϊκή υποστήριξη για τη δημιουργία υποδομών θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες εναλλακτική σταθμή, φόρτιση ηλεκτρικών αιχμάτων κτλ. Με ρωτήσατε αν αυτό θα ενταχθεί στις αναλύσεις αναχώρα, σε, αυτές, σε αυτά τα δελτία που ε, προετοιμάζουμε για την κάθε χώρα. Ναι, είναι η απάντηση γιατί θεωρούμε ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της Ενεργειακής Ένωσης. Θα δούμε και πώς προχωρούμε με τις μεταφορές ή με την ε, απαλλαγή από τις ε, εκπομπές άνθρακα στον τομέα αυτό. 18 Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί μια μεγάλη διάσκεψη για την απαλλαγή των ε, οδικών μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα και θα ήθελα το feedback ε, των εμπλεκομένων φορέων να το αξιοποιήσουμε. Θα καλέσω και άλλους επιτρόπους από την οικογένεια της Ενεργικής Ένωσης για να συζητήσουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο για να εφαρμόσουμε και να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες αυτές στην κοινή νομοθετική πρόταση. Θα γίνει και αυτή η συνάντηση λοιπόν για την απαλλαγή από τις τις εκπομπές πριν από τις θερινές διακοπές. Επίσης, θα προχωρήσουμε με το σχεδιασμό της αναθεώρησης του κανονισμού για τα πρότυπα των εκπομπών σε φορτηγά και αυτοκίνητο γήματα προβλέπεται για το 2016-2017. Χρειάζεται βέβαια προπαρασκευαστικό έργο, χρειάζονται αναλύσεις. Εργαζόμαστε επίσης και για την εκπόνηση ενός βασικού σχεδίου ε, για ένα ε, συνεκτικό κεφίες των μεταφορών για να αποφύγουμε τις συμφορήσεις. Βλέπετε τι ποτηλιάρισμα υπάρχει όταν κανείς έρχεται από το Στρασβούργο, έρχεται από την Βρυξέλλη Στρασβούρο το αντίστροφο. Θέλουμε να χρησιμοποιούν τις αστικές, ευφυείς αστικές συγκοινωνίες οι συμπολίτε μας γιατί αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλη εξοικονόμηση χρόνου και περιορισμό των ε, κυκλοφοριακών ε, συμφορήσεων. Ξέρετε επίσης ότι συζητούμε το ETS, ε, τις μεταφορές που θεωρήσαμε ότι πρέπει να ενταχθεί σε μια πρόταση που δεν αφορά το ETS. Έχουμε και τις ε, θαλάσσιες μεταφορές και τη αεροπορία. Ο ΑΙΚΑΟ θα μας βοηθήσει να διατυπώσουμε τι προτάσει μα. Θα υπάρξει ένα πολύ καλό συντονισμό, Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε στον τομέα τη απαλλαγή από τι εκπομπέ άφρακα. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε πολλά αν προωθήσουμε τεχνολογίε φιλοπεριβαλλοντικέ και ευφυές σίγουρα στο πλαίσιο και τη στρατηγική για τη θέρμανση και την ψήξη. Θα δείτε ότι θα μας απασχολήσει αυτό το ζήτημα, θα ανοίξουμε όλους τους φακέλους και, το, και για το, τη δέσμη μέτρων για τις ανώσιμες πηγές ενέργειας τις ε, ανακοινώσεις και προπαρασκευαστικό έργο για την ε, ενεργειακή απόδοση. Όλες αυτές τις προτάσεις θέλουμε να τις υποβάλουμε εντός του 2016. Τον κύριο Ντάνκαν, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση να επισκεφθώ τη Σκοτία. Έχω ε, επισκεφθεί τη χώρα αρκετές φορές, με τα χαράς να ξαναπάω τι πρέπει να δούμε. Πρέπει να δούμε τις ιδιαιτερότητες των χωρών, να τις λάβουμε υπόψη. Αλλά έχουμε και ένα κοινό στόχο που είναι μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στην Ενεργειακή Ένωση και τις ενεργειακές πολιτικές. Γι' αυτό και θα πρέπει να έχουμε ένα ισχυρό ευρωπαϊκό πλαίσιο. Πρέπει να φροντίσουμε ότι στα βασικά αυτά στοιχεία συνεργαζόμαστε, αναζητούμε ευρωπαϊκές λύσεις ή περιφερειακές λύσεις. Πιστεύω λοιπόν ή μάλλον να πω ότι η πρώτη μου αντίδραση τι επαφέ που είχαμε τα κράτη-μέλη αντιλαμβάνομαι ότι αποτελεί πρόκληση, αλλά τα κράτη-μέλη συνειδητοποιούν ότι αν ε, συγκεντρώσουν τις προσπάθειε τους ε, σε αυτή την ε, σημαντική ενεργική μετάβαση μπορούν να αποκομίσουν περισσότερα ωφέλη. Η κυρία Μαρτίν αναφέρθηκε στην ενεργική παινία, τι μπορούμε να κάνουμε για να μειώσουμε τι τιμέ της ενέργειας. Σίγουρα καλύτερη προσέγγιση είναι να φροντίσουμε να υπάρχει περισσότερο ανταγωνισμό στην αγορά ώστε οι καταναλωτές, οι πολίτες να έχουν ε, τη δύναμη και την δυνατότητα να επιλέγουν για το σπίτι τους από ποιον θα αγοράσουν ενέργεια, πώς θα την ε, καταναλώσουν, να εφαρμόσουν πιο ευφύς τεχνολογίες, ευφύ δίκτυα, τα οποία ξέρουμε ότι μειώνουν το κόστος διανομής. Και αν αυτό δεν αρκεί και αν εξακολουθούν να παραμένουν υψηλέ τιμές ενέργειας για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού, τότε σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι θα πρέπει να αναζητήσουμε τις καλύτερες δυνατές λύσεις μέσω των κοινωνικών πολιτικών κοινωνική, μεμονωμένη κοινωνική βοήθεια ή κοινωνικά τιμολόγια που ξέρετε ότι ισχύουν σε κάποια κράτη-μέλη. Διότι συμφωνώ μαζί σα ότι αν υπάρχουν τόσα εκατομμύρια πολιτών που δεν μπορούν να πληρώσουν το ρεύμα είναι κάτι απαράδεκτο και αυτό πρέπει να μα απασχολήσει και να το αντιμετωπίσουμε και ω Ευρωπαίοι αλλά και σε εθνικό επίπεδο να το δούμε ω ένα εθνικό κοινωνικό ε, πρόβλημα νομίζω ότι σας απάντησα σε εσά όταν μίλησα για την απαλλαγή από τι εκπομπέ άνθρακα προς την κυρία Ντέλη, αλλά σε ό,τι αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές υπάρχουν κάποιες ε, επιβλαβείς για το περιβάλλον ε, κρατικές ενισχύσεις. Θέλουμε λοιπόν να ισχύσουν οι προτάσεις μας και να τηρηθούν ε, τα μέτρα. Σε ό,τι αφορά τώρα την ενεργειακή εξάρτηση Ρωσία-Βόρεια Αφρική. Νομίζω ότι θα παραμείνει ε, θα παραμείνουν οι περιοχές αυτές σημαντικοί προμηθευτές ενέργειας για την Ευρώπη. Μπορούμε όμως να κάνουμε πολλά για να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από αυτές τις ε, χώρες πια. Θα έχουμε το νέο αέρα από την ε, περιοχή της Κασπίας, μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και μέσω του προγράμματος για την ενεργειακή απόδοση, θα χρησιμοποιήσουμε χώριες πηγές περισσότερο, όπως είναι η ηλιακή και η αιωλική ενέργεια και επίσης θα στεραστούμε ή μάλλον θα εργαστούμε σκληρά για να έχουμε και μια ε, πάρα πολύ καλή ενεργική στρατηγική για να αξιοποιήσουμε τις νέες ε, εξελίξεις στην αγορά. Για το πετρέλαιο ξέρουμε που είναι ένα παγκόσμιο αγαθό ότι τις τελευταίες εβδομάδες είδαμε και ότι έχει μειωθεί και η τιμή του εγραρίου σε σχέση με την τιμή του αερίου. Είναι ένα νέο φαινόμενο, θα πρέπει να το μελετήσουμε. Πρέπει να παίξουμε σωστά τα χαρτιά μας στον τομέα της ενέργειας. Άρα πρέπει να έχουμε ένα ε, ισορροπημένο εφοδιασμό. Να μην εξαρτώμαστε υπερβολικά από ε, κάποιες συγκεκριμένε χώρες όπως ε, συμβαίνει ή συνέβη για συγκεκριμένε χώρες και γενικά για την Ευρωπαϊκή Ένωση και επί σειρά ετών. Σε ό,τι αφορά το σχιστολιθικό αέριο κατάσταση στην Ευρώπη και στις, ε, είναι διαφορετική από ό,τι στις ΗΠΑ. Είναι διαφορετική η γεωλογική κατάσταση και τελείως διαφορετική αντιμετώπιση της κοινή γνώμης για την δρορμάτωση, το φράκινγκ. Εξού και θεωρώ ότι η προσέγγιση που θα λέει ότι κάθε κράτος μέλος θα πρέπει να αποφασίσει ξεχωριστά αν θέλει ή όχι να χρησιμοποιήσει αυτή την τεχνολογία. Όμως υπό την προϋπόθεση ότι θα χρησιμοποιούνται πλέον πρόσφατες ε, τεχνολογίες ε, και δεδομένα είναι κάτι εξίσου σημαντικό. Νομίζω ότι για τους Ευρωπαίους το περιβάλλον η αποδοχή αυτής της τεχνολογίας από την κοινή γνώμη είναι τελείως διαφορετική σε σχέση με τη ΣΥΠΑ. Και αυτό πολύ απλά πρέπει να το λάβουμε υπόψη. Αν είναι να χρησιμοποιήσουμε, να βασιστούμε περισσότερο σε αυτές τις τεχνολογίες, νομίζω ότι μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πιστεύω όμως, όπως είπα, ότι τα ευφύ δίκτυα θα μπορούσε να είναι το αντίστοιχο, ο αντίστοιχος ευρωπαϊκός σχιστόλιθος, αν θέλετε. Γιατί αν αναπτύξουμε και εξοπλίσουμε την τεχνολογία που ήδη έχουμε στην Ευρώπη, μπορούμε να εξοικονομήσουμε μεγάλο μέρος ενέργειας, να τη διανύμουμε με πολύ πιο αποτελεσματικό τρόπο και να περιορίσουμε κατά πολύ τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα, συμβάλλοντα και σε καλύτερε τιμέ και σε ένα πιο υγιέ περιβάλλον στην Ευρώπη. Κύριε Πέτρελε, θέλω να σας ευχαριστήσω για την, πρόστα, για την πρότασή σας. Είπατε και ο ίδιος ότι είναι τεχνική. Θα ήθελα λοιπόν να αντιλάβω και γραπτός για να τη μελετήσω ενδελεχέστερα σε ό,τι αφορά πιο πράσινες πολιτικές, πολιτικές για την ενεργειακή απόδοση. Ουσιαστικά εντάσσουμε στον προπολισμό της Ένωσης τις πολιτικές αυτές. Συνοχή. Όλα τα κονδύλια του προπολογισμού. Θέλουμε να υπάρχει ένα 20% του προπολογισμού το οποίο θα στοχεύει στην υποστήριξη πράσινων οικολογικών πολιτικών και μέτρων και θα δούμε πώς οι δικές σας προτάσεις συνάδουν με τις δικές μας πολιτικές για την ανάπτυξη της υπαίθρου όπως τις έχουμε ήδη ε, την κυρία Γκούτελαντ, για το πρόγραμμα επενδύσεων Juncker. Η ενεργειακή απόδοση είναι σαφώς ένας από τους τομείς όπου αναμένεται να υπάρξει υποστήριξη Θεωρούμε σημαντικό να υποβληθούν καλά έργα που θα περάσουν τη διαδικασία της πρώτης διαλογής, την προεπιλογή και θα χρηματοδοτηθούν δεόντως. Αυτό είναι προτεραιότητα για πολλούς δήμους, για πολλούς δημάρχους που γνωρίζω ότι έχουν έργα και θέλουν να τα στηρίξει το Ταμείο Επενδύσεων Juncker. Από κοινού και με τις τράπεζες των κρατών μελών ώστε να ομαδοποιηθούν τα αιτήματα και να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με αυτό το μέτρο για την ευφύ χρηματοδότηση. Νομίζω ότι υπάρχει μεγάλη όρεξη για τέτοιο είδους project. Η κυρία Σουίτσα, να σας πω ότι η ενέργεια στο ΚΕΡΚ είναι στρατηγική σημασία σε ένα project με το οποίο μπορούμε στην Αδριατική να προωθήσουμε τις προτάσεις μας ε, θα έχουμε αυτά τα λεγόμενα 14 1 σχέδια διασύνδεσης και στην Κροατία έχουμε τον Ιούλιο μία συνεδρία αυτής της ομάδας της ε, αρμόδιας και αν υπάρξουν κατάλληλες προϋποθέσεις για τις χώρες περιοχής και τις χώρες ενεργικής κοινότητας που δεν είναι δηλαδή μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ανήκουν στην ενεργειακή κοινότητα να έχουμε λοιπόν εξελίξεις για να αντιμετωπιστεί η υπερβολική εξάρτηση. Το κύριο Γκριπ το κάλυψα νομίζω το θέμα. Πρέπει να σεβαστούμε την κυριαρχία του ενεργειακού μείγματος, αλλά έχουμε κοινά πλαίσια ευρωπαϊκά και συμφωνίες. Στην περίπτωση της Πολωνίας τον Οκτώβριο του 2013 είχαμε την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ελήφθη μια απόφαση που νομίζω ότι σέβεται αυτή τη διαφορετική αφετηρία και νομίζω ότι αστιάζει στο συσχέσει αυτές τις τεχνολογίες για την συγκράτηση του άνθρακα κτλ. Μόλις αυτές τις τεχνολογίες νομίζω ότι θα έχουμε σημαντικά επιτέγματα, σημαντική πρόοδο στον τομέα αυτό. Σε ό,τι αφορά τη διαφορά με την Gazprom, φυσικά αρμόδιος για αυτό το θέμα ε, δεν είμαι εγώ, αλλά η συνάδελφος Μάργκρετ Βεστάγκερ και γνωρίζω ότι μέχρι στιγμής είναι θετική αντίδραση της Γκάσπρομ σε αυτή την έρευνα ε, την αντιμονοπολιακή πολιτική, υπάρχει μια επαφή με την Κομισιόν και θα δούμε τι θα γίνει. Θα υποβάλει τα επιχείρηματά της η Γκάσπρομ απαντώντας στην Κομισιόν και θα δούμε σε τι συμπεράσματα μπορούμε να καταλήξουμε. Τον κύριο Μπέλετ. Ο κύριο Μπέλετ μίλησε για την μεταρρύθμιση του συστήματο ETS, για την εμπορία εκπομπών και με των εκπομπών. Γνωρίζετε κύριε Μπέλετ πολύ καλά το θέμα. Ξέρετε λοιπόν ότι σε ό,τι αφορά την αναδιανομή των εσόδων από του πληστηριασμού, το σχέδιο είναι να σεβαστούμε τι διαφορετικέ αφετηρίε, όπω είπα, των κρατών μελών στην Ευρώπη. Το 90% λοιπόν των εσόδων θα διατεθούν σε όλα τα κράτη-μέλη και το 10% σε αυτά με το χαμηλότερο εισόδημα για να στηριχθεί η πρόοδος και ο εξυγχρονισμός των τεχνολογιών στις χώρες αυτές. Θα υπάρξει και το λεγόμενο Ταμείο καινοτομία. και έχω και το Ταμείο Εξυγχρονισμού για παροχημένους ε, ε παλαιούς ε, σταθμούς, ε, μονάδες παραγωγής ενέργειας που θέλουμε να εξυγχρονιστούν για να μην εκπέμπουν αυτές τις επιβλαβείς εκπομπές άνθρακα και να μπορούν να χρησιμοποιήσουν ταχύστα τις νέες τεχνολογίες στον αγαπητό συμπατριώτη μου τώρα να του πω ότι σε ό,τι αφορά αυτές τις κοινέ προσπάθειες που γίνεται μια μελέτη ε, για την κοινή αγορά αερίου και είπατε σωστά ότι πρέπει να είναι θελωτικό αυτό το σχήμα να χρησιμοποιείται σε περίπτωση κρίσης αλλά θα έχουμε τα αποτελέσματα της μελέτης ε, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο και θα σας ενημερώσω βέβαια ευχαρίστως ε, πιο αναλυτικά τότε για το πώς θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε τα πορίσματα της μελέτης στις μελλοντικές μας προτάσεις και σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας και την ενεργειακή απόδοση Αυτή είναι τομεί που θα τους συμπεριλάβουμε στις νομοθετικές μας προτάσεις. Μίλησα επανειλημμένως για αυτή την νομοθετική πρόταση. Νομίζω ότι θα βρούμε καλές λύσεις για το πώς θα αυξήσουμε τον, την ανταγωνιστικότητα και τον ανταγωνισμό, πώς θα μειώσουμε τις τιμές με πίεση στην αγορά, μεγαλύτερη ενεργειακή απόδοση, ένα καλύτερο, ένα πιο πρόσφορο έδαφος. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε που μου δώσατε τη δυνατότητα να απαντήσω όλα αυτά τα ερωτήματα των μελών της Επιτροπής σας. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σας, αλλά κυρίως ε, και για τον πολύ συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο απαντήσατε σε όλα τα ερωτήματα που υπέβαλαν τα μέλη της Επιτροπής μας. Νομίζω ότι μπορούμε να ολοκληρώσουμε τώρα αυτό το κομμάτι της ε, συνεδρίασής μας, ε, λέγοντας ότι η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει 29 Μαΐου στις Βρυξέλλες. 26 Μαΐου συγγνώμη, στις Βρυξέλλες. Commission and Vice President Και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.